E, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε τις εργασίες μας. Έχω ένα άσχημο νέο. η δολοφονία του Jean Serge Γάλλου αστυνομικού από την ΕΤΑ. Το πρόβλημα της τρομοκρατίας δεν έχει λυθεί. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια εκ μέρους όλου του Κοινοβουλίου στην οικογένεια του αστυνομικού. Ελπίζω να βρεθούν και οι δολοφόνοι αλλά και οι εντολή της δολοφονίας. Επίσης, άλλο άσχημο νέο, στην Κούβα συνελήφθησαν 30 διαδήλωτες ε, της ομάδας ε, Woman in White πρόκειται για μητέρες και συζύγους ε, μελών της αντιπολίτευσης που κρατούνται. Αυτές οι γυναίκες έχουν βραβευθεί με το βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς τις υποστηρίζουμε αυτές τις γενναίες γυναίκες. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση για δύο εκθέσεις. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κατάσταση του ευρώ. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Τσικλούνα και την έκθεση Σβεν Γκίγκολτ για την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ευρώ και των δημοσιονομικών το 2009. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Έντουαρτ Σικλούνα. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια ήταν, αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως θεματοφύλακα της ε, νομισματικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Στην ε, ετήσια έκθεση με αυτό το πνεύμα γράφτηκε. Βασίζεται στην ανταπόκριση προς την κρίση της ΕΚΤ και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ οικονομιών χωρών μελών. Τέλος, αντιμετωπίζονται και θέματα για τις ευθύνες που φέρει. Η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν χειρότερη από τη δεκαετία του 30 μετά από μια θετική περίοδο ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες μέλη υπέστησαν τρομερή ζημιά στις οικονομίες τους και με πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία, επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία μάλλον. Η ανάπτυξη ήταν μόνο 0,7% και η μείωση 4%. Έχει προβλεφθεί δε και για το μέλλον μία ανισομερής και χαμηλή ανάπτυξη μέχρι και το 2011. Οι περισσότερες χώρες μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλο έλλειμμα και οι προβλέψεις της Κομισιόν από το 2009 προέβλεπαν ελλείμματα των προϋπολογισμών κατά μέσο όρο 6,4%. Η αριθμή αυτή δεν πρόκειται να βελτιωθούν πολύ και φέτος. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να διορθωθούν τα πράγματα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Νομίζω ότι η ΕΚΤ έχει ανταποκριθεί σχετικά καλά προς την κρίση αυτήν. Κύριος ρόλος της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. και παρά το ότι είχαν ξεπεραστεί τα ανώτατα όρια που είχε καθορίσει η ίδια γιατί είχαν φτάσει το 4% ο πληθωρισμός τη θασεύτηκε. μέχρι να φτάσει στο 1% κατά μέσο όρο τώρα. Έκανε ό,τι μπορούσε δηλαδή για να προωθήσει την αναθέρμανση χρησιμοποίησε καινοτόμα μέτρα χωρίς τα οποία για τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πολλά από αυτά που φύλασαν τις οικονομίες των πολιτών θα είχαν καταρρεύσει. Θα μπορούσε κανείς βέβαια να πει ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ δεν μειώθηκαν τόσο πολύ όσο τα αμερικανικά. Και οι ενέσεις χρημάτων από την έκτη σε πολλά ιδρύματα δεν ωφέλησαν και τους πελάτες τους, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η οικονομική αναθέρμανση. Πολλές τράπεζες μάλιστα χρησιμοποίησαν τις ενέσεις αυτές για να βελτιώσουν τη δική τους μόνο κατάσταση και συνέχισαν να πληρώνουν πριν στους υπαλλήλου των. Η αντιμετώπιση των, της κρίσης αυτής φυσικά είναι κάτι που πρέπει να, ε, προς το οποίο πρέπει να αντιδράσουμε στεναρά και είμαι σίγουρος ότι και οι συνάδελφοι θα το αναφέρουν. Πιστεύω ότι ο διάλογος μεταξύ ΕΚΤ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το επικοδομητικό και που αναπτύσσεται θετικά. Πρέπει να συνεχιστεί και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί στενότερα τους διορισμούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μεταξύ των οποίων και, ο προσεχής και τον προσεχή της Πρόεδρο σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και για την έγκριση ή το διορισμό του νέου αντιπροέδρου της. Η ΕΚΤ είναι υπόλογη προς τους πολίτες της Ευρώπης μέσω ακριβώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Πάνω απ' όλα η κρίση έχει αποδείξει ότι οι αγορές αν δεν διευθετηθούν δεν αυτοδιορθώνονται πάντοτε. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε και να συμπληρώσουμε τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί, ιδιαίτερα δε την, να υποστηρίξουμε την ίδρυση ενός μιας ειδική υπηρεσίας παρακολούθησης κρίσεων ώστε να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση. Μου έχει δοθεί ένα πρόσθετο λεπτό κύριε Πρόεδρε. Όχι δεν σας έχει δοθεί. Επόμενος συζητητής είναι ο κύριος Σβέν Γκίγκολντ. Ορίστε. κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά συντάχθηκε σε μια στιγμή στην οποία έχουμε μια τεράστια πρόκληση για την Ευρωζώνη. Δεν έχει περάσει αυτή η στιγμή. Η οικονομική κατάσταση ανησυχεί τους πολίτες και εμάς ακριβώς τώρα συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων σε πολύ καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αυτή η έκθεση και θα ήθελα λοιπόν να σας την παρουσιάσω. Είναι σαφές πως ε, και με την έκθεση της ε, Κομισιόν και με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου που θα έρθουν στην Ολομέλεια βλέπουμε ξεκάθαρα πως αφενός πρέπει να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση, αφετέρου η κρίση η οποία σταθεροποιήθηκε κάπως, ε, υπάρχει κάποια ανάπτυξη μέχρι να περάσει σε μια δεύτερη φάση βεβαίως σημαίνει τεράστια ελλείμματα και χρέη που είναι το τίμημα για να βγούμε από την κρίση αυτή. Το μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές. Πρέπει γρήγορα να επανέλθουμε στον ορθό δρόμο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα χρέη στα παιδιά μας. Από την άλλη όμως είναι εξίσου σαφές πως η σταθερότητα από μόνη της δεν αρκίζει. Η Ευρώπη θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα. Λείπουν αυτά τα μέτρα ειδικά όσον αφορά τις ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης και θα πρέπει να ενισχυθεί και ο δημοσιονομικός συντονισμός όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό ακριβώς οι υπεύθυνοι πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα και αυτό σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν ο καθένας από τη μεριά του να επιμένει στα εθνικά προνόμια και ωφέλη που έχει και αυτό ισχύει ακριβώς όσον αφορά την ευθύνη της Κομισιόν και του Eurogroup. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Τι προτείνουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα αποτελεσματικά μέτρα οικονομικού συντονισμού. Δεύτερον, η διαρθρωτική εξάρτηση της Ευρωζώνης από κάποιους πόρους να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν να εξαρτώμεθα συνεχώς από τις ε, τιμές ε, πετρελαίου και λοιπόν φυσικών πόρων. Τρίτον, δεν θα πρέπει απλά να ρυθμιστούν αποτελεσματικά οι αγορές μετά από αυτήν την κρίση, αλλά κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν λογικές προτάσεις για αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει. Τέταρτον, δεν είναι δυνατόν να κινούμαστε ενάντια στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο στόχος εδώ πέρα δεν ήταν η κοινωνική συνοχή. Και αυτό υποβαθμίζεται ακριβώς επειδή κάποια κράτη-μέλη πληρώνουν τεράστια επιτόκια για να χρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ευρωομόλογα, να επιδειχθεί κάποια αλληλεγγύη για να βοηθήσουμε αυτά στα κράτη-μέλη. Επίση, οι απαραίτητε διορθώσει που πρέπει να γίνουν στην πολιτική, τη δημοσιονομική, δεν μπορεί να είναι ει βάρο τη αγοραστική δύναμη του λαού. Και ένα τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι η αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα τη φορολογία. Η Κομισιόν επιτέλου πρέπει γρήγορα να καταθέσει προτάσει για ένα, μια κοινή φορολογητέα ύλη όσον αφορά τις επιχειρήσεις. και να υπάρξουν επίσης όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις μια έκθεση αναχώρα στην οποία δραστηριοποιούνται και ακριβώς όσον αφορά τη συνεργασία του κυρίου Μόντι και για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς έχει μεγαλύτερη σημασία η φορολογική συνεργασία πρέπει να δοθεί προβάδισμα σε αυτήν και όχι στο φορολογικό ανταγωνισμό έτσι μόνο εάν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε στα παιδιά μας χρέη αλλά μια ευρωζώνη η οποία θα ε, συνεργάζεται και δεν θα έχουμε ένα ανταγωνισμό προς τα κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ζαν Κλοντ Τρισέ. Έχετε τον λόγο κύριε πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι για την συζήτηση σχετικά με την έκθεση του 2008 για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με βάση τα όσα έγιναν πέρυσι νομίζω πως η φετινή συζήτηση είναι σαφώς εντονότερη αλλά αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα να μπω στην επικαιρότητα. Όπως ξέρετε Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ε, στενές σχέσεις που έχει με το Κοινοβούλιο που ξεπερνούν τα όρια που έχουν οριστεί από τις συνθήκες. και οι δύο εξαιρετικές εκθέσεις που ακούσαμε καταμαρτυρούν του λόγου του αληθές. Εγώ θα σας αναφέρω την πολιτική που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις νομισματικές ε, λύσεις. Ε, θα σας πω τι σκοπεύουμε να κάνουμε και θα σας πω και τι γίνεται με την τωρινή κατάσταση. Πρώτα για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Το 2009 η ΕΚΤ λειτουργούσε όπως ε, λέει ο κύριος Σικλούνα σε ένα περιβάλλον που οι ιστορικοί θα περιγράψουν ως το πιο δύσκολο για τις ανεπτυγμένες οικονομίες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μετά την ένταση της οικονομικής ε, κρίσης ε, το 2009 ξεκίνησε με συγχρονισμένη ελεύθερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίας. Μέχρι τον περσινό Απρίλιο έπεφτε μήνα με το μήνα η οικονομική δραστηριότητα. Κατά την περίοδο αυτή, αυτό το οποίο ήταν σημαντικό για να διατηρήσουμε την ε, εμπιστοσύνη ήταν η ικανότητα να λάβουμε τα άμεσα και εξαιρετικά εκείνα έκτακτα μέτρα που ήταν αναγκαία ενώ ταυτόχρονα παραμέναμε σταθεροί στην προσήλωσή μας στην ε, σταθερότητα των τιμών. Επίσης είχαμε και τα έκτακτα μέτρα τα οποία είναι γνωστά συλλογικά ως μια ενισχυμένη στήριξη βοήθησαν την Ευρωζώνη και τη λειτουργία της αγοράς χρήματος με αποτέλεσμα να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες δανεισμού και πίστοσης της πραγματικής οικονομίας καλύτερης από ό,τι θα γινόταν μόνο με μια πολιτική επιτοκίων. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό και μέσω των επιτοκίων της ΕΚΤ για τον δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Βασική μας αρχή είναι να επιστρέψουμε στα φυσιολογικά επίπεδα καθώς εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση θα αλλάξει η συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά. Γι' αυτό το Δεκέμβριο του 2009 αρχίσαμε σταδιακά να αποσύρουμε κάποιο από τα έκτακτα μέτρα ρευστότητα που είχαμε λάβει με βάση τη βελτίωση των χρηματαγορών. Δηλαδή μειώσαμε τον αριθμό και την συχνότητα και την οριμότητα των μέτρων αναχρηματοδοτήσεως. Επίσης στηρίζαμε την ρευστότητα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ρευστότητα τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο φέτος. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, η νομισματική μας πολιτική αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη και η πολιτική που ακολουθούμε θα οφείλει στην σταθερότητα των τιμών πρόθεσμα Να αναφερθώ τώρα σε κάποια από τα ζητήματα που αναφέρονται στο ψήφισμα και στην έκθεση. Για ζητήματα υπευθυνότητα ε, λογοδοσίας και διαφάνειας εκτιμούμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το επικοδομητικό του πνεύμα. Καλωσορίζω λοιπόν την συνεχή στήριξη της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων για τον τριμηνίο διάλογό μας. Όπως είπε και ο εισηγητής, εμείς δίνουμε λόγο στον Ευρωπαίο πολίτη, κατά το οποίο πρακτικά σημαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε πως η ΕΚΤ είναι μία από τις πιο διαφανείς παγκόσμια κεντρικές τράπεζες μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Νομισματικής ναι. Πολιτικής δίνουμε συνέντευξη τύπου κάτι το οποίο ε, να θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλε μεγάλες τράπεζε Επίσης δημοσιεύουμε και τα πρακτικά μας για να εξηγηθεί και η λογική μας. Όπως ξέρετε έχουμε εντείνει τις επικοινωνιακέ μας προσπάθειες για να εξομαλυνθεί η αντίδραση των χρηματαγορών, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και να μπουν τα θεμέλια της ανάκαμψης. Επίσης ζητήσατε τις απόψεις μας για να υπάρξει ένα μέσο στο οποίο θα γίνεται η εκαθάριση μέσων όπως τα credit default swaps, η συμφωνίες συνταλλαγής κινδύνου. Όπως σας είπα, η στόχοι μας είναι γνωστοί και το να υπάρξει μια κεντρική εκαθάριση αντισυμβαλωμένων είναι πάρα πολύ σημαντική για να μειωθούν και η υπερβολικοί κίνδυνοι και να είναι σε καλύτερη θέση εξαγωγής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει κατάχρηση για κερδοσκοπία. Θα πρέπει λοιπόν οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να ερευνούν τυχόν απρεπείς συμπεριφορές. Και εδώ πέρα νομίζω πως συμφωνούμε απόλυτα με το Κοινοβούλιο. Να πω τώρα κάποια πράγματα για την ΩΝΕ σε καιρούς δύσκολους. Υπάρχει μια ανάκαμψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η κρίση τελείωσε. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε πως ο ρυθμός της ανάκαμψης θα είναι άνισος και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και οπισθοχωρήσεις. Από την άλλη αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς ε, θα πρέπει τα ιδρύματα αυτά να παίξουν επικοδομητικό ρόλο και η λιδία αλήθως θα είναι το κατά πόσον θα εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία για να διασφαλιστεί αυτός ο ρόλος θα πρέπει να λειτουργεί και να ε, εξετάσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στον τραπεζικό τομέα. Επίσης έχουν γίνει και θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι τράπεζες και για το πώς λειτουργούν οι χρηματαγορές. Πρέπει να επινοήσουμε μηχανισμούς και κίνητρα για να διασφαλίσουμε πως ε, δεν θα ξεφύγει με καταστροφικό τρόπο, δεν θα ξεφύγουν οι χρήματα με καταστροφικό τρόπο όπω έγινε ακριβώ πριν την κρίση. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιε είναι αυτέ οι συστημικές διαταραχέ που δημιουργούν οικονομικέ δυσκολίε για του λαού τη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, το οποίο εξετάζει, εξετάζει αυτή τη στιγμή τη σχετική νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και συνδέονται με τα δημόσια οικονομικά όπως και πάλι τόνισε ο εισηγητής ε, και αφορούν λοιπόν και το δημόσιο χρέος. Υπάρχει λοιπόν σαφής κατανομή ευθυνών. Σε σχέση με αυτή την κατανομή ευθυνών όλοι μπορούν να βασιστούν στην δέσμευση της έκτη για τη σταθερότητα των τιμών της Ευρωζώνης μεσοπρόθεσμα με βάση την τελευταία μας προβολή στο τέλος του έτους στα 12 χρόνια του ευρώ ο πληθωρισμός ε, ετήσιος μέσος όρος θα είναι 1,95% σύμφωνα δηλαδή με τον ορισμό μας περί σταθερότητας που είναι γύρω στο 2%. Η στρατηγική της ΕΚΤ και η πολιτική που έχει ακολουθήσει είναι συνεπής. Η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ δεν αφορά μόνο την νομισματική ένωση αλλά και την οικονομική Ένωση. Τα μέτρα της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διατηρούν υγιή τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία ανταγωνιστική. Τη στιγμή αυτή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει κέρυες αποφάσεις πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η ευημερία της Ένωσης απαιτεί δράση από όλους. Η νομισματική ένωση της Ευρώπης είναι πολύ περισσότερο από κάποιες νομισματικές ρυθμίσεις είναι μια κοινή μοίρα. Θα το επαναλάβω, συμμεριζόμαστε μια κοινή μοίρα. Ε, Η μοίρα αυτή είναι για το κοινό μας καλό και ήταν το όραμα των ιδρυτών της Ένωσης. Δεν είναι θέμα ευκολία η νομισματική ένωση είναι μέρος μιας διαδικασίας ένωσης των λαών της Ευρώπης που ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιστεύω πως συχνά μειώνουμε τα επιτεύγματα της Ευρώπης και ασκούμε γρήγορα κριτική στα θεσμικά όργανα και στις διαδικασίες μας, αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργούν και σε δύσκολους καιρούς κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και οι διαδικασίες παρέμειναν αποτελεσματικέ. Δεν είχαμε τα τραυματικά εκείνα γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να εντείνουν την, Κρήτη, όπως, ε, την κρίση όπως αυτό ε, έγινε στι ΗΠΑ. Και στο πλαίσιο αυτό εκτιμώ την δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωζώνης που έγινε στο τελευταίο Συμβούλιο για να αναλάβουν συντονισμένη δράση, αν χρειάζεται αυτό, για να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Δράτω με της ευκαιρίας, κύριε Πρόεδρε, να σας επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων Δευτέρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σκοπεύει να παραμείνουμε όσον αφορά την αξιολόγησή μας σε επίπεδο 3β και έχουμε και ένα συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα προστασίας του ευρωσυστήματος. Θα σας δώσω τις τεχνικές λεπτομέρειες όταν θα σας ενημερώσω στη... για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μας στις 8 Απριλίου. Να σας πω κύριε Πρόεδρε πως η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος πριν από μία δεκαετία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο επιτεύγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερία στην Ευρώπη. Η παγκόσμια οικονομική κρίση απαιτέλεσε μια πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε και όλα τα κράτη-μέλη απέτρεψαν το να γίνει χειρότερη η κρίση με το να έχουμε και μια νομισματική κρίση όπως είχαμε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον κέριων αποφάσεων και θα πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ευημερία για να γίνει η ένωσή μας ακόμη πιο ελκυστική για να δουλεύει και να εργάζεται κανείς. Αυτό σημαίνει πως χρειαζόμαστε καλύτερη επιτήρηση όπως είπαν οι εισηγητές και καλύτερη συνεργασία και να υπάρξει ξανά μια αίσθηση κοινού στόχου όπως είχαν οι ιδρυτές μας οι οποίοι είχαν όραμα και αυτά τα οποία είδαμε τις τελευταίες μέρες ευεβεβαιώνει το πόσο στο μέλλον είχαν δει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Χαιρετίζουμε εδώ την παρουσία του Επιτρόπου που έχει και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ΕΚΤ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε την ετήσια δήλωση για την Ευρωζώνη. Κατά την προετοιμασία της γνωρίζαμε ότι τα θέματα της επικαιρότητα θα ήταν κέρια. Ίσως μάλιστα να έχουν πάρει και υπερβολική σημασία, τουλάχιστον για μένα, τελευταία. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συζητητές, Σικλούνα και Γκίγκουλτ για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις και για να σεβαστώ την ανεξαρτησία της ΕΚΤ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την δική της παρουσίαση που είναι πολύ ουσιώδη συμβολή στη συζήτησή μας για τον οικονομικό συντονισμό και την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι η εκτίμηση που δείχνουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς, τους, προς τον κύριο Γκίγκολτ ε, απορρέει από τη μεγάλη του γνώση των θεμάτων αυτών. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε ότι το ευρώ δεν είναι μόνο ένα τεχνικό νομισματικό θέμα η διευθέτηση αλλά είναι, βρίσκεται στην καρδιά του οράματος της Ευρώπης και πρέπει αυτό το κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα να το στηρίξουμε όχι μόνο τώρα αλλά και για το μέλλον στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Από το 1999 η Ευρωζώνη υπήρξε ζώνη σταθερότητας. Προφύλαξε τους πολίτες μας από τις οικονομικές διαταράξεις, αλλά από τα τέλη του 8 η Ευρωζώνη επλήγει σκληρά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και παρά τη σχετική ανάκαμψη και τα φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ασταθείς. Οι πρόσφατες τάσεις της αγοράς έδειξαν ότι η οικονομική διακυβέρνηση και η σταθερότητα ε, δεν είναι ακόμη διασφαλισμένες και αυτό φαίνεται από την Ελλάδα. Η Ελλάδα τώρα θέλει να στοχεύσει το 4% του ελλείμματος μετά από τη λήψη των σκληρών και τολμηρών μέτρων της Ελληνικής Βουλής. Αυτή τη στιγμή θα είναι ιστορική για την Ελλάδα. Αλλά Ούτε η Ελλάδα, ούτε το σύνολο της Ευρωζώνης έχουν ακόμη ανακάμψει. Γι' αυτό η Κομισιόν ενθαρρύνει τις χώρες της Ευρωζώνης να πάρουν μια πολιτική απόφαση, ένα μηχανισμό για να διασφαλίσουν την σταθερότητα στη ζώνη αυτή. Ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί άμεσα ανάλογα με τις ανάγκες σύμφωνα και με αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες χωρίς αυτόματο χαρακτήρα βέβαια. Για μας σας μπορώ να σας διασφαλίσω ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη και διατεθειμένη να δημιουργήσει και να συντονίσει ένα τέτοιο όργανο η υπηρεσία που να χρησιμοποιείται μόνο εάν τα χρειάζεται. Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα μέλη της Ευρωζώνης και την ΕΚΤ για να βρεθεί μια τέτοια λύση και που θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας. Τώρα για την άμεση διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης πρέπει να αναλύσουμε πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Η ελληνική κρίση έχει δείξει ότι υπάρχει ανάγκη για ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση πράγμα το οποίο αναγνωρίστηκε και στην, ως νομική βάση τέθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό προετοιμάζουμε προτάσεις για την εφαρμογή του άρθρου 136 της συνθήκης και η Κομισιόν θα τις υποβάλει προτάσεις για ενισχυμένη οικονομική συνεργασία δηλαδή και ενισχυμένη επιτήρηση της οικονομικής συμπεριφοράς των χωρών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συζητητής Γκίγκολτ στο σημείο 28 του ψηφίσματος του εκφράζει τη λύπη του γιατί δεν ανελήφθησαν δεσμευτικά μέτρα και υποσχέσεις από τις κυβερνήσεις για να ενισχυθεί η Ευρωζώνη και είπε ότι χρειάζεται μια πιο στεναρή αντιμετώπιση για να βρεθεί μια λύση. Καταρχάς πρέπει να αποφευχθεί η αύξηση των ελλημάτων και άρα χρειάζεται καλύτερη επιτήρηση των, της συμπεριφοράς των χωρών της Ευρωζώνης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε δεσμευτικές και αυστηρές συστάσεις προς τις χώρες και υπολογίζω και στη δική σας υποστήριξη για την πρόταση αυτή. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη χρήση των υπαρχών των εργαλείων γιατί το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να κάνει συστάσεις οικονομικής πολιτικής στις χώρες μέλη εφόσον υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας. Στο παρελθόν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει πολλές φορές. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Κομισιόν έχει τώρα τη δυνατότητα να κάνει τέτοιες προειδοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 121 άμεσα σε κάποια χώρα μέλος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μπορούμε να το πράξουμε εφόσον μερικές χώρες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό να γίνεται η προειδοποίηση εγκαίρως. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επειδή πλησιάζει το τέλος του χρόνου μου, θα συνεχίσω για τις μακροοικονομικές, δεν θα αναφέρω τις μακροοικονομικές διαταράξεις, αλλά θα περάσω κατευθείαν στα συμπεράσματά μου. Εγώ συμμερίζω με τις απόψεις των εισηγητών και θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει δείξει χωρίς αμφιβολία ότι η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι το δεδομένο. Ίσως να έχουμε ξεπεράσει τη χειρότερη ήδη φάση, αλλά η ανάπτυξη είναι ακόμη ευαίσθητη, δεν είναι διασφαλισμένη. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, δηλαδή την αποφυγή των ελλημάτων. Τα δύο χρόνια της κρίσης, όσα αφορολογικά μέτρα και να ελήφθησαν, έχουν εξαλείψει σχεδόν τα αποτελέσματα μιας εικοσαετίας οικονομικής ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα σύννεφα θα σκεπάζουν για πολλά χρόνια την, το οικονομικό τοπίο της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αναθέρμανση και γι' αυτό είναι καιρός να ληφθούν εξαιρετικά μέτρα και σημαντικές αλαβαθμιές αλλαγές για την διασφάλιση της πλήρους απασχόλησης ή πληρέστερης απασχόλησης. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων τώρα θα μιλήσουν πρώτα το ΕΛΚ η κυρία Σοφία Ικονή για τρία ολόκληρα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκίγκολτ που μας έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολτ. Η έκθεσή του είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ετήσια δήλωση της Κομισιόν για την Ευρωζώνη και τα δημοσιονομικά και συμπεριλαμβάνει και πολύ χρήσιμες προτάσεις. Βέβαια χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση, την περσινή οικονομική κρίση που ήταν η χειρότερη που γνώρισε η Ένωση από την ίδρυσή της. Δύο διδάγματα έχω βγάλει από αυτή την έκθεση. Πρώτον, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει δείξει ότι είναι κάτι το θετικό και το ευρώ, σταθερό και κοινό νόμισμα έπαιξε το ρόλο πραγματικά μιας ασπίδας προστασίας της Ευρωζώνης και επέτρεψε σε πολλές χώρες να αποφύγουν υποτίμηση του εθνικού τους νομίσματος που θα είχε χειροτερέψει την κρίση. Η Ευρωζώνη λοιπόν έγινε ακόμη πιο ελκυστική για τους υπόλοιπους όπως φαίνεται από την Ισλανδία. Η ενεργή και ευέλικτη στρατηγική της ΕΚΤ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την διατήρηση της δραστηριότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη οικοδομήθηκε από κρίσει, αλλά εδώ φάνηκε ότι η οικονομική Ευρώπη είναι και αποτελεσματική και απαραίτητη. Αυτό είναι το δεύτερο δίδαγμα που εξάγω. Να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση πανενοσιακώς. Διότι η μόνη πραγματική οικονομική ευρωπαϊκή πολιτική είναι η νομισματική. Ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών είναι περιορισμένος, ενώ η Ευρωζώνη που όπως λέει και η έκθεση στοχεύει στην ολοκλήρωση όλων των οικονομιών της Ένωσης πρέπει να διαθέτει και μία αποτελεσματική διακυβέρνηση για όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς της. Καταρχήν μακροοικονομική και δημοσιονομική επιτήρηση την οποία επεξεργαζόμαστε τώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να γίνει με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να είναι ένα πραγματικό εργαλείο συντονισμού, δημοσιονομικού συντονισμού. Σε τέτοιες περιόδους κρίσης η σημαντική μείωση των εισοδημάτων και τα κίνητρα που έχουν δοθεί ως μέτρα για σταθεροποίηση των οικονομικών παραγόντων και παραμέτρων είναι απαραίτητη. Η μείωση του ελλείμματος και του χρέους είναι κάτι βασικό διότι αφορά το μέλλον των παιδιών μας Πρέπει όμως να επιδείξουμε και κάποια πνεύμα καινοτομία να εφεύρουμε καινούριε νέες δημοσιονομικές πολιτικές και προγράμματα, ώστε να υπάρξει μια πραγματική ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα εξ ονόματος των σοσιαλιστών ο κύριος Χονκόκ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση του Σβεν Γίγολτ είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τωρινό πλαίσιο. Πόσο μάλλον πιο εύστοχη αυτή η έκθεση, διότι ο βουλευτής είναι Γερμανός και θέλει να επιστήσει την προσοχή των Ευρωπαίων για τα στρεβλά για τις στρεβλές επιπτώσεις της πίεσης των μισθών στη Γερμανία. Δηλαδή οι Γερμανοί οδηγούν όλη την Ευρώπη σε, μία, σε ένα μισθολογικό αποπληθωρισμό ιδιαίτερα σημαντικό. Και οι χώρες οι οποίες έχουν ένα τρέχον ισοζύγιο ελληματικό και εφόσον δεν μπορούν να υποτιμήσουν μειώνουν την κοινωνική προστασία και μειώνουν τους μισθούς. Έχουμε λοιπόν καθυστέρηση, εσωτερική οικονομική καθυστέρηση και αρνητική ανάπτυξη, αρνητικό δίκτυο ανάπτυξης ακόμη πριν ξεσπάσει η κρίση της ρευστότητας. Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνεται το χρέος. Έχουμε λοιπόν μια γενική χρηματοπιστωτική απορρίθμιση στην Ισπανία, στην Ιρλανδία που τη διαπιστώσαμε με την κρίση των subprimes. Ακούγοντας αγαπητοί συνάδελφοι την συζήτηση Πολλοί βουλευτές προσπαθούν να ξεχάσουν τα διδάγματα αυτής της κρίσης. Μα η κρίση δεν βρίσκεται πίσω μας. Η κρίση υπάρχει και στο βαθμό που δεν λαμβάνονται μέτρα για την αλάφρυνση της μισθολογικής πίεσης και καλούνται τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πολιτικές λιτότητας οι οποίες θα σκοτώσουν οποιαδήποτε εγγενέσει την ανάπτυξη και πουθενά δεν θα λυθεί το πρόβλημα ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ισπανία ούτε αλλού διότι δεν θα υπάρχουν φορολογικά έσοδα και δεν θα καλυφθούν τα ελλείμματα. Το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι αρνούνται να αναιρέσουν τη θέση τους για τις μισθολογικές πιέσεις. Αλλά πιστεύω ότι η έκθεση του Σβέν Γκίγκολτ είναι, πολύ, είναι χρήσιμη διότι βάζει το πρόβλημα και το συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Ραμόν Τρεμόζα Ιμπαλσές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Σικλούνα, ο οποίος είναι μέγας γνώστης των κεντρικών τραπεζών, και τον κύριο Γκίγκολτ. Με... Συζητήσαμε πολύ και καταφέραμε να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ δεν θα μιλήσω για το ευρώ. Εγώ καινούριο είμαι στην πολιτική. Και μέχρι πριν από 9 μήνες δίδασκα μακροοικονομία στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Εγώ ζούσα το 2008 για ακαδαμικούς λόγους με την οικογένειά μου στο Λονδίνο και έβλεπα αυτήν την τρομερή πτώση της ε, στερλίνας 30% σε λίγες εβδομάδες. Και όλοι οι Εγγλέζοι συνάδελφοί μου φτώχυναν απότομα με την πτώση της, της στερλίνας. Σκεφτείτε τι θα γινόταν και για μας λοιπόν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο για το ευρώ. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι το ευρώ αποτελεί ένα αγκυροβόλι σταθερότητας. Δεν φτώχυναν οι πολίτες της Ευρώπης με το ευρώ. Ήταν ένα σίγουρο λιμάνι το ευρώ. Σε όλες αυτές ε, τις ε, νομισματικές τρικυμίες. Και ο καθηγητής ε, Μάρτς, ο οποίος ήταν ευρωσκεπτικιστής, δημοσίευσε ένα βιβλίο πριν από κανένα χρόνο όπου επενεί τελικά το ευρώ. Δεν βρίσκεται σε κρίση το ευρώ. Οι φορολογικές κρίσεις ορισμένων κρατών μελών δημιουργούν δυσκολίες στο νόμισμα. Το ευρώ το θαυμάζουν οι οικονομικές ελίτε της Ινδίας, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ρωσίας. Δεν είναι ρίσκο για τις μεσογειακές οικονομίες είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης των οικονομιών τους στις καλές πρακτικές, τις προθυμένες και ρεφορμιστικές καλές πρακτικές των κέντρων των χωρών της ε, Βόρειας Ευρώπης. Η τεχνητή υποτίμηση του κινέζικου νομίσματος συνέβαλε στη δημιουργία της κρίσης στη ζώνη του ευρώ δεν θα πρέπει εμείς να επιβαρύνουμε τις χώρες που είναι οι πιο εξαγωγικές. Η οικονομική ιστορία διδάσκει ότι η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών. Η Γερμανία θα πρέπει να ενισχύσει την κατανάλωση στη χώρα και να αποτελέσει κινητήρα για την ανάπτυξη όλης της, επόμενης, όλης της Ευρώπης. Εγώ είμαι καταλανός βουλευτής, έρχομαι από την Καταλωνία που συμμετέχει με το 28% στις συνολικές εξαγωγές των, της Ισπανίας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να επιβαρύνουμε τους καλύτερους. Το ευρώ έχει ιδιαίτερο πρεστίζ παγκοσμίω. Θα πρέπει όμως να έχει και γύρω του και μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει να δημοσιεύονται οι διάλογοι και τα πρακτικά γύρω από το ευρώ, όπως κάνουν και οι άλλες μεγάλες τράπεζες. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους Φιλίπ Λαμπέρ. Ήθελα να μιλήσω γαλλικά, αλλά επειδή θέλω να με καταλάβει και ο Επίτροπος Ρέιν θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σημερινή κατάσταση και να δούμε το μέλλον. Έχουμε τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία, σας το λέω, δεν τα υποστηρίζουν οι πράσινοι. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως έχουμε ήδη τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. 16% των Ευρωπαίων κάτω από το όριο της φτώχειας δεν είναι μικρό νούμερο. 40% των νέων Ισπανών κάτω των 25 άνεργοι δεν είναι μικρό νούμερο και θα μπορούσα να συνεχίσω. Και μετά μας λείπουν και οι πόροι, κλιματική αλλαγή κτλ. Όλα αυτά σημαίνουν πως χρειάζονται επενδύσεις στις ε, υποδομές, ε, την εκπαίδευση, έρευνα κτλ. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε ταχύτητα. Ο κύριος Φαν μετά την σύνοδο του Φεβρουαρίου είπε πως χρειάζεται καλύτερο συντονισμός μακροοικονομικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως όσον αφορά τα έξοδα του προϋπολογισμού χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο εκ των προτέρων και ελεγχομοτήτων. Η Ελλάδα έχει μια αεροπορία τόσο μεγάλη όσο τη Λουθβάφε. 4% του ΑΕΠ πάει στρατιωτικές δαπάνες. Είναι μια μικρή, μια μικρή χώρα και οπλίζεται σαν να μην υπάρχει αύριο αλλά αν δούμε μόνο τις δαπάνες δεν θα επιτύχουμε. Πρέπει να συντονίσουμε τα φορολογικά έσοδα. Γιατί πρέπει τα φορολογικά έσοδα να μην είναι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από το κεφάλαιο. Να είναι κεφαλαιοχικά έσοδα, να υπάρξει πραγματική συνεισφορά των εταιριών, όχι μόνο στα χαρτιά, αυτό που είχαμε πει δηλαδή οι πολυεθνικές να αναφέρονται αναχώρα. Επίσης φόρος άνθρακα και να αλλάξουν οι συμπεριφορές για να βρωθούν εισοδήματα. Και αυτό δεν γίνεται με το να ζητάμε από τις χώρες να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Θέμε περισσότερη ολοκλήρωση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, οι κυβερνήσεις μας θα αποδειχθούν ανίκανες το, για να ισορροπήσουν τους προπολογισμού και να έχουν ταυτόχρονα ικανοποιήσει τι κοινωνικές ανάγκες και να κάνουν επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι η Ευρώπη. Η επιλογή είναι μεταξύ ενός ψηλότερου βαθμού ολοκλήρωση, όχι μόνο συντονισμού, και παρακμής. Τα διδάγματα της Κοπενχάγη δεν είναι μόνο ότι χάσαμε τη συμφωνία, είναι πω η Ευρώπη πλέον δεν έχει σημασία γιατί συντονιζόμαστε μεταξύ μας εμείς εδώ πέρα και δεν δρούμε. Αυτή είναι η συνεισφορά μας σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κέιν Σουίμπορν, εξ ονόματος των συντηρητικών. Ευχαριστώ. Επειδή δεν προέρχομαι από χώρα της Ευρωζώνης, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά που θα σας πω θα τα προσέξουν οι συνάδελφοι. Τα προβλήματα της κρίσης ας τα λύσουν τα μέλη της Ευρωζώνης. Παρ' όλα αυτά και εμείς επηρεαζόμαστε από την κρίση φυσικά. Κατά τις καλές εποχές γνωρίζαμε ορισμένες μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων που σήμερα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Βέβαια η Γερμανία δεν έχει το ίδιο έλλειμμα με την Ελλάδα, αλλά έχουν αλλάξει κυρίως, πρέπει να παρατηρήσω, οι νοοτροπίες ως προς την αποταμίευση παραδείγματος χάρη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαφορετική φορολογική πολιτική, αλλά χρειάστηκε και εκείνο να μπλοκάρει πολλές δραστηριότητες στο δημόσιο τομέα και για μας λοιπόν έχουν περάσει πια οι εποχές των παχιών, παχαίων αγελάδων. Δεν είναι αλήθεια βέβαια για κανέναν μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη ότι οι κυβερνήσεις μπορούν πια μαγικά να λύσουν τα νομισματικά προβλήματα και η Γερμανία το αναγνωρίζει κατά το πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία είχε κάνει μεγάλες δημόσιες δαπάνες και γι' αυτό σήμερα είναι σε πιο ισχυρή θέση. Ο δημόσιος τομέας έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει κατά την κρίση στηρίχθηκε ο τραπεζικός τομέας και τώρα πρέπει να ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα να δώσει τα χρήματα που χρειάζονται για, το για τα υπόλοιπα μέτρα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων επιχειρηματιών παραδείγματο χάρη και αυτό είναι βασικό στοιχείο για την διατήρηση του ιδιωτικού τομέα. Όσες χώρες εφάρμοσαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η δική μου, και η δική μου πολιτική που δεν μπορούσε να στηριχθεί, τώρα υποφέρουν περισσότερο από την κρίση. Ευχαριστούμε. Νικόλαος Σαλαβράκος. Jürgen Α, όχι, Κλούτερ, Κλούτερ. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, λειτουργεί το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δράτω με τις ευκαιρίες ε, να επανέλθω στην Ελλάδα, γιατί θεωρώ πως η κρίση στην Ελλάδα μας ε, δίνει χρήσιμες πληροφορίες και για την ε, κατάσταση της Ευρώς. Πρώτα απ' όλα έχουμε την παρατήρηση της κυρίας Ευρώ ότι θα μπορούσε στην ανάγκη να διώξει την Ελλάδα από το ευρώ. Η ομάδα μου η το θεωρεί κάτι τέτοιο παράλογο. Από τη μία μιλάμε για κοινή μας μοίρα και από την άλλη στην πρώτη μεγάλη δυσκολία λέμε να βγάλουμε μια χώρα έξω. Αναξιοπρεπές. Κυρίως όμως αυτό θα ήταν δήλωση χρεοκοπίας για, την, για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Γιατί λέμε πως το ευρώ είναι η ελπίδα μας για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και τώρα λέμε πως πρέπει να αποκλείσουμε από αυτό την Ελλάδα. Και τώρα βλέπουμε πώς ακολουθεί η επόμενη χώρα. Η Πορτογαλία υποβαθμίστηκε χτες όσον αφορά την ε, πιστοληπτική της ε, ικανότητα και πώς θα εξηγήσουμε στους εργαζόμενους ότι αυτοί πρέπει να πληρώσουν αλλά από την άλλη τα φορολογικά τους χρήματα στηρίζουν τις τράπεζες. Όποιος δρά έτσι πολύ απλά διακινδυνεύει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλη την δίκαια κριτική κατά της Ελλάδας και οι σύντροφοι από την ε, Ελλάδα βλέπουν πως πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά παρόλη την κριτική η κρίση δεν είναι ευθύνη της ε, Ελλάδας. Υπενθυμίζω εδώ πέρα τις αποφάσεις ε, της Ευρωζώνης που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ευρώ δεν προσφέρει απάντηση στην διαφορετική ανταγωνιστικότητα των ε, χωρών. Αντί να εξάγει όπως η Γερμανία, η Ελλάδα γονάτισε. Οπότε η κρίση είναι και κρίση της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης. Γι' αυτό και τελειώνω, ζητούμε απαγόρευση να αρθεί η απαγόρευση της ε, οικονομικής ε, σύνδρομης κρατών μελών θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, κοινά ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως ε, κάνει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και να απαγορευθούν credit default swaps. Ναι, τελειώνω. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θα αναλάβω εγώ τώρα την Προεδρία. Ο επόμενος ομιλητής λοιπόν για ένα λεπτό είναι ο κύριος Σαλαβράκος. Η 25 Μαρτίου είναι γενέθλια μέρα της Ευρώπης και της Ελλάδας. Στις 25 Μαρτίου του 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης ανέτειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 25 Μαρτίου του 1821 γεννήθηκε η Ελλάδα. Σήμερα, στη γενέθλια μέρα τους, δοκιμάζονται και η Ευρώπη και η Ελλάδα. Η Ευρώπη στη συνοχή της και η Ελλάδα στα οικονομικά της όλοι στην αίθουσα αυτή γνωρίζουμε ότι από τις 15 χώρες της Ευρωζώνης οι 6 έχουν υψηλό δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα. Όλοι στην αίθουσα αυτή γνωρίζουμε ότι και οι 30 χώρες μέλη του ΟΣΑ έχουν χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ και κατά 30% υψηλότερο ένα του 2008 οι ίδιες οι Ηνωμένε Πολιτείε σε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση που ζούμε προσπαθούν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα τυπώνοντας κυρίως χαρτονόμισμα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Ελλάδα έλαβε αυστηρά οικονομικά μέτρα λιτότητας μέχρι της εξαντλήσεως των πολιτών τους. Πολλοί θα πούν ότι καλά να πάθει η Ελλάδα και να πληρώσουν τα, τα σφαλματά της. Ναι, κάποιοι θα λογοδοτήσουν γι' αυτό. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι η ελλάδα εισάγει προϊόντα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από τη γερμανία κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι εξάγει. Παρακαλώ λοιπόν να ληφθεί υπόψη από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η αντιμετώπιση των κερδοσκόπων θα δημιουργήσει γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη πολιτική. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να, να σέβεστε το χρόνο. Λοιπόν, θέλουμε να, να ψηφίσουμε κιόλα κάποια στιγμή και εντάξει πρέπει να τηρείτε κάποια στιγμή ο χρόνος των ομιλητών. Ναι, έχετε, έχετε δίκιο. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε τον χρόνο. Ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν σας βγάζω το καπέλο για αυτό το οποίο κάνατε τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αισθάνεστε πως αυτή την στιγμή εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων φοβούνται πως ε, το τι θα γίνει με το ευρώ. Πρώτα απ' όλα έχουμε βεβαίως τα πακέτα αυτά, τα έκτατα τα οποία λάβατε για την αναχρηματοδότηση της ρευστότητα. Αλλά βεβαίως υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος του πληθωρισμού και ειδικά ως Αυστριακός σας προειδοποιώ για το τι ε, θα γίνει όσον αφορά και εμάς και την Γερμανία. Προσέξτε, δεν μπορεί να τιμωρηθεί η χώρα αυτή η οποία παρήχε τη μεγαλύτερη σταθερότητα λόγω άλλων οι οποίοι ξόδευαν αλόγιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπάλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως ισχυώδης ηγητής του ΕΛΚ για την ε, έκθεση για την ΕΚΤ είμαστε ικανοποιημένοι. Είχαμε και καλή συνεργασία και με τον κύριο Σικλούνα και τον κύριο Τριμούσα για την ισορροπημένη αυτή έκθεση για το 2008. Ο πρόεδρος ο κύριος Τρισέ και ο συμφωνούν μαζί μας. Νομίζω πως το πρώτο έτος της κρίσης το 2008 ήταν πάρα πολύ δύσκολο και με βάση αυτή την πρόκληση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανταποκρίθηκε σε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει και έδρασε σωστά. Ε, νομίζω πως η έκθεση Σικλούνα το αντικατοπτρίζει αυτό και θεωρώ επίσης πως η κατάσταση της έκθεσης δεν είναι καθόλου απλή και στο προσεχές μέλλον θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη. Πρώτα απ' όλα η κρίση δεν έχει περάσει ακόμα και βεβαίως πέραν των ρυθμιστικών μέτρων ανακύπτουν και νέες προκλήσεις και προβλήματα για την ΕΝΚΤ. Νομίζω λοιπόν πως είναι σημαντικό η τράπεζα προσεχώς να συνεχίσει να φροντίζει για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης να ακολουθήσετε λοιπόν και να παραμείνετε στην καλή πορεία που έχετε χαράξει από την άλλη κύριε Τρισέ το είπαμε αυτό και στον πολιτικό διάλογο που είχαμε να διατηρηθεί και η πολιτική ανεξαρτησία της τράπεζας ακριβώς ε, όσον αφορά και την μελλοντική σας σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Καθώς βεβαίως θα εμπλακείτε εντονότατα και ως ε, πρόεδρος της ε, ΕΚΤ. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει οι διαβουλεύσει αυτού του Συμβουλίου να αποτελέσουν κριτήριο των αποφάσεων της ε, Τράπεζας και νομίζω πως θα πρέπει να συνεργαστούμε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζάνι Πιτέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, κύριε Επίτροπε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Η κατάσταση έχει ήδη περιγραφεί. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θεραπευτική αγωγή. Και το πρώτο σημείο θα είναι η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση που χωρίς αυτήν το οικονομικό σύστημα δεν θα μεγαλώσει και το χρέος θα γίνει αβάστακτο. Η Ελλάδα πρέπει να, να εξορκιστεί, πρέπει να την εξορκίσουμε ούτως ώστε να μην έχουμε το εφέ όπου θα πέσουν όλες οι χώρες από το βάρος του χρέους. Πολιτική για την Ελλάδα λοιπόν, οικονομικά μέσα στη διάθεσή μας για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και μία πολιτική για τη διαχείριση του κατεπήγοντος. Εγώ άκουσα σήμερα το πρωί τοποθετήσεις οι οποίες επενούν τις δόξες του ευρώ. Αλλά γιατί να μην φανταστούμε το ευρώ όχι μόνο το ευρώ ως ένα νόμισμα που μας σώζει από τον πληθωρισμό αλλά ως ένα νόμισμα που με ένα μικρό χρέος μας επιτρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ρευστότητα μέσα από τα ευρωμόλογα. Εγώ συμφωνώ στην ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και θέλω να πω συμπερασματικά συνάδελφοι και θέλω να το πω καθαρά και εξάστερα σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται απλά και μόνο να επιπλέουμε. Δεν χρειάζεται μία δειλή Ευρώπη. Ντόνα Μπόντιο λέει ο μιλητής μιλώντας για τους προμεσείς πόζοι. Χρειάζεται μία θαραλέα Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπόουλς έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρισέ, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Είχαμε μία δύσκολη εβδομάδα στην Επιτροπή με τους Προέδρους της ΕΚΤ και του ε, Eurogroup και τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Τράπεζας. Συμφωνούμε όλοι πως χρειάζεται ισχυρότερη επιτήρηση των κρατών μελών με σωστά στατιστικά στοιχεία για να μπορεί να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Ξεκίνησε ήδη η σχετική δουλειά με περισσότερες εξουσίες για την Eurostat και η Επιτροπή αναμένει να παίξει και αυτή τον αυξημένο ρόλο της. Υπάρχουν όμως και άλλα κριτήρια, άλλοι δείκτες που πρέπει να γίνουν σεβαστοί, καθώς ο μεγαλύτερος συντονισμός για να οδηγηθούμε σε μακρονομική σταθερότητα είναι μια επιλογή, αλλά τη δοκιμάσαμε. Θυμηθείτε τι είχε γίνει το 2001 για την προειδοποίηση του ΕΚΟΦΗΝ στην Ιρλανδία επί καιρό πλεονασμάτων. Οπότε γνωρίζουμε τα μαθήματα. Το να έχουμε πειθαρχία σε καιρού πλεονασμάτων είναι ακόμη δυσκολότερο από ότι σε καιρό ελλημάτων. Και όπως ακριβώς δεν το έκαναν αυτό οι χρηματαγορές οδηγούμαστε σε κρίσεις. Όσον αφορά δε τις ανισορροπίες μεταξύ κρατών μελών πρέπει να δούμε πού χάνεται η ανταγωνιστικότητα, πού συχνά πάει χέρι με χέρι με το να σέρνουμε τα πόδια μας στην κοινή αγορά και με το να μην γίνονται μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές όπως στις συντάξεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει αυτομάτως έλλειμμα. Και τέλος όπως είπε και ο κύριος Σικλούνα η ρυφστότητα που παρέχει η ΕΚΤ ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο στην κρίση αλλά δεν πέρασε στην πραγματική οικονομία. Συχνά επανεπενδύθηκε σε άλλα μέσα που απέδιδαν περισσότερο σε τόκους. Και εδώ πέρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπωσδήποτε κάπου κάποιοι αυτό το θεωρούν ότι αξίζει και μπόνους. Οπότε θα πρέπει να ακούμε τις εκκλήσεις τέτοιων τραπεζών όσον αφορά την ε, καθυστέρηση επιβολής των κανόνων ε, κεφαλαϊκής επάρκειας. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν τον λόγο έχει ο κύριος Τρεμόπουλος για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι πρόκειται για μια σημαντική έκθεση ε, η οποία αποτελεί και έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό ε, των τάσεων που υπάρχουν ε, στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. εντοπίζει στοιχεία κοινωνικής συνοχής που δεν παρουσιάζονταν σε ανάλογες συζητήσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. θα θέλαμε να σηματοδοτεί και μια σημαντική στροφή και τη πολιτική τη ευρωπαϊκής Ένωση συνολικότερα. βέβαια αναφέρεται στο 2009 ενώ στο 2010 είχαμε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν φυσικά και την ελλάδα τη χώρα μου. αυτό που θα μπορούσε να βγάλει κανείς ως συμπέρασμα είναι ότι πέρα από την ε, νομισματική ένωση χρειάζεται όπως λένε και πολλοί άλλοι και οικονομική και πολιτική ένωση και το ευρώ θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα μίνιμουμ δίχτυ κοινωνική ασφαλείας αυτό για την κοινωνική συνοχή. αυτό προκύπτει και από τα διάφορα που λέγονται για την ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό είναι ανακριβή. Όπως για παράδειγμα δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι η παραγωγικότητα της Ελλάδας δεν ήταν πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Eurostat για το 2007 και το 2008 ήταν περίπου γύρω στο 90%. Η αύξηση του ελλείμματος του υπροπολογισμού και του δημοσίου χρέους τα τελευταία δύο τρία χρόνια στην ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης των εσόδων της μείωσης ε, των εσόδων από το εξωτερικό όπως από τον τουρισμό και την ναυτιλία λόγω της κρίσης αλλά και της αύξησης των δημοσίων δαπανών φυσικά και υπάρχουν ε, ε, σπατάλες αλλά και προσλήψεις στο δημόσιο με διάφορες μορφές. σίγουρα όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν και να ζητήσουμε και αυτό το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και να μην αρκούμαστε σε εκκλήσεις γενικόλογες να μην θυγούν πολύ τα χαμηλά εισοδήματα. θα πρέπει να γίνει έλεγχος των δαπανών και των εξοπλισμών αλλά και αυτών που αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως όμως των εσόδων που μειώθηκαν επίσης σημαντικά. δεν θα πρέπει να μειωθούν ε, τα εισοδήματα των ε, μεγάλων τμήματων του πληθυσμού που είναι στο όριο της φτώχειας. προφανώς αυτά είναι ζητήματα που αφορούν και την ε, ε, σύνοδο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα εδώ στις βρυξέλλες όμως σηματοδοτεί ή θα πρέπει η έκθεση giegold θα πρέπει να σηματοδοτεί και μια γενικότερη αλλαγή και ενσωμάτωση των θέσεων αυτών στο σύμφωνο σταθερότητα. πάνω απ' όλα δεν χρειάζεται καμιά προσφυγή στην απαράδεκτη πολιτική του διεθνού νομισματικού ταμείου όπου κοντά στα άλλα έχει και ένα έλλειμμα βιωσιμότητα. ευχαριστώ. Σωστά αναφέρθηκαν οι κύριοι Ρεν και Τρεις στη σημερινή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση της Ελλάδας και η λύση κατά την άποψή μου είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέρα με τη μέρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρώ πως το δούνο του είναι ο σωστός οργανισμός για να βοηθήσει την Ελλάδα και όσοι δεν μπορούν να τηρήσουν επίσης τους κανόνες του παιχνιδιού θα πρέπει ίσως να σταματήσουν να παίζουν το παιχνίδι. Να δούμε την κατάσταση. Η ε, Ελλάδα όταν μπήκε στο ευρώ συμπεριφέρθηκε σαν το ματίο των δελφών. Τα νούμερα ήταν τελείως ομιχλώδη. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τιρμορούνται οι άλλες χώρες του ευρώ γιατί θεωρούνται συνυπεύθυνε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό συγκεκριμένα ερωτώ τους κυρίους Τρισέ και Ρεν. Γνωρίζετε το ότι τα νούμερα τα οποία έδωσε η Ελλάδα όταν μπήκε στο ευρώ δεν ήταν σωστά και πλήρη. Και αν όχι, δεν θα έπρεπε να το ξέρατε. Αυτή την απάντηση αναμένω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φαντάλεν, για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ στους συμπατριώτες μου ό,τι καλύτερο για την 25η Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε, η καπιταλιστική κρίση έχει σαν αποτέλεσμα την ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων ταυτόχρονα έδωσε στο κεφάλαιο την ευκαιρία να εντείνει την εφαρμογή των αντεργατικών επιλογών. υπό το κράτο τρομοκράτη των εργαζομένων η πλουτοκρατία ξεκίνησε έναν πραγματικό πόλεμο ενάντια σε θεμελιώδη μισθολογικά και κοινωνικά δικαιώματα με στόχο την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. βασικό πυλώνα τη αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσει των κρατών μελών είναι η ΕΚΤ. η σκληρή πολιτική που ασκεί έχει αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. η από την ίδρυσή τη συνεχεί εκκλήσει για συμπίεση των μισθών και επιτάχυνση των καπιταλιστικών διαρθρώσεων βρήκαν πρόσφορο έδαφο στην καπιταλιστική κρίση. Η ΕΚΤ στάθηκε ουσιαστικό αρρωγό τη προσπάθεια τη πλουτοκρατία να ρίξει το βάρο τη κρίση στου ώμου των εργαζομένων. Διοχέτευσε περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ στι τράπεζε και στου μονοπωλιακού ομίλου. Σήμερα όμω καλεί του εργαζόμενου αυτοί να πληρώσουν τα σπασμένα και να επιστρέψουν αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό χρειάζεται ενδυνάμωση του αντιυμπεριαλιστικού αγώνα, τη πάλη για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη πάλι για τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία, τη πάλι για τον σοσιαλισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αγγουράκη. Ο κύριε Μπλουμ. Uh, uh, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, φαίνεται ότι εγώ ζω σε άλλο σύμπαν όταν μιλάτε για τις επιτυχίες του ευρώ. Για να προσγειωθούμε λίγο ανεργία των νέων στην Ιβυρική Χερσόνησο και σε πολλές χώρες είναι χρόνια κατάσταση. 30-40%. Καμία σχέση με την κρίση. Καταστροφή. ΑΕΠ κατά κεφαλήν στη ΣΥΠΑ. Πολύ πιο μπροστά από μας. Ανάπτυξη στις χώρες του Ειρηνικού. Πολύ πιο μπροστά από μας. Οπότε το ευρώ δεν είναι επιτυχία. Ήδη είναι αποτυχία καταραίει μπροστά στα μάτια μας. Ας δούμε τα βασικά. Δεν υπάρχει δανειστής τελευταίας καταφυγής. Εξού και η ελληνική κρίση και η πορτογαλική που έρχεται. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο σε μια διαχείριση ενός νομίσματος. Είτε είναι ιδανική η ζώνη του νομίσματος, είτε όχι. Δεν υπάρχει συντονισμός δημοσιονομικής πολιτικής. Οπότε είναι καταδικασμένη η υπόθεση να αποτύχει και αποτυγχάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και δημιουργούν πλούτο και οι υπόλοιποι που ξοδεύουν τον πλούτο. Οι πολιτικοί δηλαδή και οι γραφειοκράτες. Και είμαστε πάρα πολύ τέτοιοι. Εμείς είμαστε στο σβέρκο των άλλων. Έχουμε καθίσει. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τα έξω αλλιώς η κατάσταση θα γίνει μόνο χειρότερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κορνιλία Βαντίμ Τιδόρ. Microphone, please. Excuse me, sir. Doamnelor și domnilor, cauza majoră a crizei este mafia. Am să vă dau câteva Λοιπόν, η κρίση είναι μαφία και να σας δώσω και παραδείγματα για την Ρουμανία. Και τα λέω αυτά γιατί τα ξέρω. Να σας δώσω παραδείγματα αυτά. Από το 90 και μετά, 6.000 επιχειρήσεις ιδιωτικοποιήθηκαν της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί μόνο το 1% 7 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση απλώς έγινε πέρασμα ιδιοκτησίας χωρίς πώληση. Πρόκειται λοιπόν για οικονομία της ζούγκλας και όχι για οικονομία της αγοράς. Έτσι γίνεται στα Βαλκάνια. Η τοπική μαφία ε, η τοπική μαφία συνεταιρίστηκε με τη διεθνή μαφία. Πρόκειται λοιπόν για τη δαποθήκη από την Ελλάδα ως και αλλού. Εμείς ε, κάναμε εξαγωγή της επανάστασης στον προηγούμενο αιώνα. Τώρα τι κάνουμε εξαγωγή της πτώχευσης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν την διαφθορά και να εξαφανίσουμε τους διεφθαρμένους. Η κατάσταση της διαφθοράς είναι τρομερή και άμα δεν σταματήσουν οι απαταιωνίες στις χώρες μας τότε θα πέσει η Ευρώπη σαν χάρτινος πύργος. Χρειάζονται ριζικές λύσεις. Η μαφία πρέπει να θαυτεί, όχι να ελέγχεται. Ο Βέργεν Λάγκεν. Κύριε Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαν Κλωτρισέ για τα τελευταία 6 χρόνια που ήταν πολύ επιτυχής και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το, τους για την έκθεσή του. Και κύριε Ρεν, έχετε τώρα δύσκολα μπροστά σας και ελπίζω η Κομισιόν επιτέλους να έχει το θάρρος να κάνει μια πρόταση για να συμπληρώσει το ελιπές σύμφωνο σταθερότητας. Δεν μπορεί να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση από τους υπουργού Οικονομικών γιατί αυτοί ακριβώς απέτυχαν. Πρέπει να εισαχθεί μεγαλύτερος αυτοματισμός. Δεν θέλουμε οικονομική διακυβέρνηση από τους υπουργού. Χρειαζόμαστε αυτόματη αντίδραση όταν υπάρχουν παραβιάσεις και βοήθεια υπό την ηγεσία της ΕΚΤ και της Κομισιόν. Και θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρόεδρος για την ε, Ευρωζώνη. Χαιρετίζω το ότι είπατε πως χρειαζόμαστε παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και το ζήτημα δεν είναι να ανταγωνίζεται η μία ε, χώρα της Ευρωζώνης στην άλλη, αλλά την Ασία και τη ΣΥΠΑ. Δεύτερον, πως το ότι χάρη στις πλεονασματικές χώρες ε, έχει ισορροπημένα ε, βιβλία η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το εκτιμήσει αλλιώ Θα ήταν πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Και πρέπει οι χώρες να εξάγουν. Πρέπει να αναπτυχθούν. Τέλος, όσον αφορά την Γερμανία, το πώς η Γερμανία κατάφερε στο εσωτερικό της ε, να γίνει πιο ενιαία είναι παράδειγμα και για τους άλλους. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι δυνατόν όμως να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα οποία έπρεπε να τιμωρούνται και να επιβραβεύονται αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν τα σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει πολλή δουλειά μπροστά της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ η κυρία Άννη Ποδηματά τώρα για δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους ε, δύο εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Σε λίγο ξεκινούν ε, οι εργασίες μιας από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής και η πολυφωνία εξακολουθεί να μένεται γύρω από το λεγόμενο ελληνικό ζήτημα και γύρω από το αν και κατά πόσο θα προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα λειτουργεί σε περίπτωση ανάγκης ως δίχτυ προστασίας για την οικονομία που θα έχει ανάγκη και για τη σταθερότητα της ευρωζώνης συνολικά. είναι αναμφισβήτητο ότι η βασική ευθύνη για αυτή την κατάσταση ανήκει στην ελλάδα και την έχει αναλάβει πλήρως. υπάρχουν όμως και άλλες ευθύνες συλλογικές. το κοινό νόμισμα πρόσφερε πολλά αλλά έχει και σημαντικές αδυναμίες. στα έντεκα χρόνια λειτουργίας της ονε δεν θέλαμε να δούμε και να αναγνωρίσουμε ότι το χάσμα ανταγωνιστικότητας και οι σημαντικές ανισότητες και ανισορροπίες ανάμεσα στις οικονομίες της ευρωζώνης δεν είναι συμβατές ούτε με τη βιωσιμότητα ούτε με τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. οι κερδοσκοπικές επιθέσεις που μέχρι τώρα αφορούν κυρίως την ελλάδα αλλά να που μόλις προχθές οδήγησαν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πορτογαλίας και έχουν ήδη στραφεί σε βάρος άλλων χωρών όπως ιταλία η ισπανία χωρίς κανείς να ξέρει ποια θα είναι η συνέχεια το έχουν καταστήσει σαφές. εάν λοιπόν θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε προς ένα νέο μοντέλο ενισχυμένου οικονομικού συντονισμού και οικονομικής διακυβέρνησης που θα σέβεται αγαπητέ συνάδελφε κύριε langen τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και παράλληλα όμως θα μπορέσει να προχωρήσει πέρα από το στενά νοούμενο δημοσιονομικό συντονισμό σε έναν οικονομικό συντονισμό με επιπρόσθετα κριτήρια την κάλυψη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την αηφόρο ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρισέ, κύριε Επίτροπε. Το ευρώ νομίζω πέρασε τις, τις εξετάσεις, αν και υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, αλλά είμαι σίγουρος πως κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα για μια ευρωπαϊκή λύση, αν και μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα είπε ο κύριος Τρισέ. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα τρομακτικά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδείχθηκε βράχος στους δημοσιονομικούς τυφώνες. Βράχος σταθερότητας και για χώρες και εκτός της Ευρωζώνης. Το ευρώ εγγύθηκε την σταθερότητα και ήταν η προϋπόθεση για την δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σημαντικών σε ε, καιρούς δύσκολους. Ε. Τώρα για την ε, Ελλάδα. Τι κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη αν δεν υπήρχε το ευρώ. Τα ελλείμματα υπήρχαν πάντα και βεβαίως ε, αυτό ε, δεν θα βοηθούνταν με υποτιμήσεις ε, τις οποίες είχαμε ζήσει και εμείς στο παρελθόν και δεν βοηθούν ήμουν και εγώ σε ανάλογες επιτροπές στην Σουηδία πρέπει τα ελλείμματα να είναι χαμηλά να υπάρχει καλύτερη επιτήρηση και καλύτερο συντονισμός της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημοσιονομικός συντονισμός ε, του προϋπολογισμού δηλαδή είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε. Επίση αναφέρθηκε η κερδοσκοπία. Αν δούμε παραδείγματο χάρη τη δική μου τη χώρα και το τι έγινε στη δεκαετία του 90 όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των ε, κερδοσκόπων ήταν θετικό το ότι εμείς λάβαμε και μπορούσαμε να λάβουμε μόνοι μας μέτρα. Γνωρίζαμε πως είχε φτάσει αυτός ο καιρός και λάβαμε τότε αυτά τα απαραίτητα σκληρά μέτρα και το ίδιο πρέπει να κάνουν και άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσαρνίτσι έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της ΕΚΤΟ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη στρατιωτική γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι προηγούμενοι. Εγώ δεν εκπροσωπώ τους τραπεζίτες εδώ πέρα, αλλά την πολιτική ομάδα της οποίας η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από χώρες της Ευρωζώνης. Επομένως, η άποψή μου ίσως είναι διαφορετική. 36 ο αριθμός ε, του Προέδρου ΣΕ, είναι ο αριθμός των βουλευτών που τον άκουσαν. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαστε τεμπέληδες. Όχι. Απλώς οι ευρωβουλευτές δεν πιστεύουν ότι η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αποτελέσει λύση για την κρίση, ότι θα αποτελέσει σωσίβιο. Ο Επίτροπος Ρεν είπε ότι το ε, Βρω είναι το σωσίβιο αλλά και την άλλη μεριά λέει ότι η Ελλάδα πλήγεται από την κρίση γιατί μπήκε πολύ νωρίς στην Ευρωζώνη σε αυτή την όαση σταθερότητας. Όλα αυτά είναι αντιφατικά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που είπαν ότι η κρίση δεν έχει περάσει. Η οικονομική κατάσταση σε πολλές χώρες είναι σαφώς αρνητική. Η ανεργία στις περισσότερες χώρες αυξάνει. Τα μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα βαθαίνουν την κρίση Κύριε Τρισέ και κύριε Ρεν, και μιλώ θεσμικά, την κρίση δεν τη βλέπατε. Είχατε τα σημάδια. Όταν ξέσπασε η κρίση, κρυφτήκατε πίσω από την αντίληψη ο καθένα να λύσει μόνο του τα προβλήματα. Τώρα ερχόσαστε και επαναλαμβάνετε μονότονα επιτήρηση των ελλημάτων, πειθαρχία στο σύμφωνο σταθερότητα. Κατά την άποψή μου το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα δεν είναι τα υγιή δημοσιονομικά. Γνωρίζετε ότι χώρε όπω η Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουν τον δανεισμό, είναι βορρά στου κερδοσκόπου, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτονται τα θεσμικά και τα πολιτικά κενά που έχει η ονε. κατόπιν τούτου θα σα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητα. η αιμονή στην εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητα ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεση είναι φανερό ότι θα ανεβάσει και θα αυξήσει τι περιφερειακέ και τι κοινωνικέ ανισότητε, θα αυξήσει την ανεργία και θα μηδενίσει κάθε αναπτυξιακή προοπτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη είναι δύσκολη. Η οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα όμως πρέπει να προέλθει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το δίνει του είναι ιδανικό για να βοηθήσει εδώ πέρα την Ελλάδα. Σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου φαίνεται πως είναι μόνο πολιτική σκέψη. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα ένα νέο όργανο εάν δεν έχουμε εξαντλήσει τους υπάρχοντες κανόνες. Δεν ξέρω εάν χρειάζεται κιόλας. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα οι κανόνε προβλέπουν κυρώσει για παραβίαση του Συμφώνου Σταθερότητα. Και θα πρέπει να λάβει η Eurostat την εντολή για έλεγχο των στοιχείων που δίνουν τα ε, κράτη-μέλη για να εφαρμοστεί έτσι ο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκέντι κατόπιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία μεγάλη έλλειψη της έκθεσης είναι ότι δεν δακτυλοδεικνύει τους ε, υπεύθυνου, υπεύθυνους, τους φταίχτες που ελπίζω κάποια στιγμή να τους πούμε με το όνομά τους. Εμείς ε, αντιμετωπίζουμε κρίση σήμερα, αλλά ποιος φταίει για την κρίση, όχι όποιος δουλεύει και πληρώνει τους φόρους του. Οι τράπεζες τη δημιούργησαν ε, την κρίση και κατακορόιδεψαν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Στην Ουγγαρία μία πολυεθνική αν θέλει να έρθει στη χώρα θα πρέπει να της δοθεί μια άδεια. Μετά προσλαμβάνει προσωπικό. Αλλά προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να, δεν έχει καν το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε. Όλες αυτές οι παρατυπίες συμβάλλουν στην κρίση. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Ο κύριος Γκαρσία Μαργάιο. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο γιατί ο κύριος Γκαρσία Μαραγκάγιο δεν είναι εδώ. Πρόεδρε, η κρίση που περνάμε είναι η χειρότερη τα τελευταία 80 χρόνια. Η ιστορία των subprimes και η πτώχευση της, ε, της Lehman Brothers οδήγησε την Ευρώπη να, έχουμε σε να έχει πάνω από 23 εκατομμύρια ανέργους και ένα τεράστιο έλλειμμα η Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε να δώσει ρευστό στο σύστημα, να κάνει ενέσεις συνεργαζόμενο με τις βασικές νομισματικές αρχές. Εμείς ε, σήμερα θέλουμε ανάκαμψη χωρίς πληθωριστικές πιέσεις και θα πρέπει να αποφύγουμε μία απόσυρση, απότιμη απόσυρση των έκτακτων μέτρων που θα υποσκάψουν την οικονομική ανάκαμψη. Πρέπει να ενισχύσουμε το νομισματικό και οικονομικό πυλώνα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις τιμές στάθερες και να μειώσουμε το γενικότερο χρέος θα πρέπει να, να σταθεροποιήσουμε τα δημοσιονομικά, θα πρέπει συντονισμένα και έξυπνα να επανενεργοποιήσουμε την οικονομία μέσα από τις επενδύσεις, από την κατανάλωση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εμείς θα πρέπει να διορθώσουμε τις ε, ε, παγκόσμιες ανισότητες εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Εμείς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε καλύτερα διεθνώς όταν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ανταγωνιστικότητα των τρεχουσών μας πληρωμών. Η Ελλάδα χρειάζεται η υποστήριξη, αποφασιστική υποστήριξη είναι το κοινό μας συμφέρον. Πρόκειται για κάτι που θα βλάψει όλους τους Ευρωπαίους. Αλληλεγγύη χρειάζεται για το ευρώ. Ε, το ευρώ δεν είναι μόνο ένα νόμισμα. Όπως το είπε και ο κύριος Τρισέ. Και θα το πω στα ελληνικά τώρα, που είναι και το... Το αύριο είναι το κοινό μας μέλλον λένε στα ελληνικά. Το ευρώ, συγγνώμη. Uh, uh, Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έπληξαν όλες τις χώρες της Ένωσης μέσα και έξω από την Ευρωζώνη. Δυστυχώς οι νέοι φέρουν το μεγαλύτερο βάρος. Τα δημοσιονομικά πολλών χωρών μελών έχουν αποδυναμωθεί από την κρίση και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, η Ιρλανδική κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα το 8 και το 9 ήδη, με στόχο να μην ξεπερνιέται το 14% του ΑΕΠ και το έλλειμμα έμεινε στο 11,6% το 2010. Η δράση της κυβέρνησης έχει αναγνωριστεί και διεθνώς από τις αγορές. Από τον περασμένο Δεκέμβριο που ενεκρίθη ο προϋπολογισμός έχουν σταθεροποιηθεί τα πράγματα. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα υπόθηκε ότι η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών με τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας επένεσε την δράση της Ιρλανδικής κυβέρνησης η οποία βρίσκεται στην πρωτοπορία σε σύγκριση με άλλες κυβερνήσεις όπως του Ηνωμένου Βασιλείου των οποίον τα ελλείμματα ξεπερνούν το 10% επίσης και πρέπει και αυτές να κάνουν προσαρμογές για να διατηρηθεί η σταθερότητα των δημοσιονομικών τους. Καταλήγω ότι η Ιρλανδία παραμένει μια καλή τοποθεσία για επενδύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεπεράσατε λίγο το χρόνο σας, ο κύριος Σμπίγνιεφ Ζιόμπρο. Η κρίση στην Ευρωζώνη μας δείχνει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να πλήξουν τα οικονομικά σχέδια και τις αρχές μας και αξίες μας. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν ορισμένες χώρες μπορούν να μπουν στην Ευρωζώνη. Το ευρώ δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σχέδιο, είναι και ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο στόχευε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτή η βιασύνη όμως μπορεί να πλήττει τους φορολογούμενους πολλών χωρών μελών. Πρέπει λοιπόν να ανασύρουμε τα σωστά διδάγματα. Το ευρώ δεν είναι απάντηση στα διαρθρωτικά προβλήματα των διαφόρων οικονομιών δεν είναι μία απάντηση στο χρέος και στο έλλειμμα. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα εκεί όπου δημιουργήθηκε. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα και τις δύο εκθέσεις και από ό,τι άκουσα σήμερα ενδυναμώθηκαν οι πεπιθήσεις μου. Εκτός από ορισμένε εξαιρέσεις πάντοτε γίνεται λόγος για λιτότητα και για το σύμφωνο σταθερότητας που δεν ανταποκρίνεται βέβαια πλέον σε τίποτα. Μπορεί όλοι μιλάνε για την οικονομική διακυβέρνηση βέβαια, αλλά εμείς θέλουμε και μια πολιτική Ευρώπη που να μπορεί να ελέγχει, να έχει επιλογές οικονομικές και κοινωνικές και να μπορεί να παρεμβαίνει. Η ελληνική κρίση ή δείχνει τι συμβαίνει. Η Γερμανία επιβάλλει τους όρους της και στις Ηνωμένε Πολιτείες η Κεντρική Τράπεζα αγόρασε κρατικά ομόλογα, άρα παρενέβη. Ενώ για την Ελλάδα πάντα οι ίδιοι πληρώνουν την ύφη. Οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, ενώ είναι τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης. Δεν είναι αυτά τα μέτρα που χρειαζόμαστε, αλλά μια άλλη Ευρώπη, οικονομική και κοινωνική, που να εξυπηρετεί τους περισσότερους και όχι μόνο τους λίγους. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Γιαροσλάβ Πάσχα. Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις για την ετήσια δήλωση της Ευρωζώνης δείχνουν πώς έχουν τα πράγματα από το 2009 η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί προφανώς και το θέμα δεν είναι να ψέξουμε με μονομένες χώρες. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις από χώρα σε χώρα και είναι διαφορετικά και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Παρά τις προσπάθειες της Ένωσης να συντονίσει τα μέτρα αντιμετώπισης και να εφαρμόσει κάποια αλληλεγγύη, είδαμε ότι ορισμένες χώρες δεν είχαν συμπεριφερθεί όπως έπρεπε και απέτυχαν. Πρέπει λοιπόν να δούμε μήπως οι διάφορες οικονομικές τίγρεις όπως η Μαλαισία και η Κίνα έχουν να επιδείξουν τίποτε καλύτερο και γιατί πρέπει στο άμεσο μέλλον να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τα δημοσιονομικά μας αλλά εκτός αυτού πρέπει να προσπαθήσουμε να αναδομήσουμε τα πράγματα, να αναδιαρθρώσουμε γιατί είναι γεγονός ότι μόνο όσοι παράγουν δημιουργούν πλούτο για τους υπόλοιπους. Κυρία Τζιόρι, Ευχαριστώ. Το το η έκτα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 ξέσπασε η οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημοσιονομική κρίση που κατέληξε σε πάγωμα των δανειοδοτήσεων. Η ΕΚΤ αντιμετώπισε άμεσα την κρίση αλλά δεν ξεχνάμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι δυστυχώς υπήρξε και κάποιο πρόβλημα για τις χώρες ιδίως που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Εδώ πρόκειται για άνηση μεταχείρισή τους, αντίθετη με το πνεύμα των συνθήκων. Η ΕΚΤ δηλαδή δεν έκανε, δεν έπραξε το καθήκον της. Δεν χορήγησε χρήματα χωρίς εγγυήσεις σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Οι Σουηδοί πήραν χρήματα χωρίς εγγυήσεις αλλά για την Πολωνία και την Ουγγαρία επιβλήθηκαν εγγυήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές αποσταθεροποιήθηκαν και οι χώρες αυτές αντιμετώπισαν ακόμη μεγαλύτερη κρίση από τις υπόλοιπες. Μιλάμε τώρα για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας αξιολόγηση των κρίσεων. Πρέπει να υπάρξει κάποια εξισορρόπηση εδώ πέρα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια άνηση μεταχείριση. Και ακόμη παραπέρα, τι θα είναι η υπηρεσία αυτή. Εδώ η ΕΚΤ πρέπει να παίξει τον κύριο ρόλο, διότι διότι λέγω εκείνη θα διευθετεί τις έρευνες και πρέπει οι χώρες της Ευρωζώνης και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην διαχείριση της υπηρεσίας αυτής. Αλέως θα υπάρξει άνηση μεταχείριση η οποία σε περιόδους κρίσης θα έχει τρομερά αποτελέσματα πρέπει να διασφαλίσουμε το πνεύμα των συνθήκων. Ευχαριστούμε. Ο Ζόρ Σαμπίν Κούτας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κεντρική ιδέα της παρουσίασης της δήλωσης για την Ευρωζώνη αφορούσε την κρίση. Καλό είναι λοιπόν νομίζω που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε χρήματα στις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης αλλά και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης επλήγησαν από την κρίση και μια παρέμβαση της ΕΚΤ προς τις χώρες αυτές θα χρειαζόταν επίσης η αύξηση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους καθώς και της ανεργίας μεταξύ ιδιαίτερα των νέων κάτω των 25 ετών είναι χαρακτηριστικά όλων των ευρωπαϊκών χωρών και το σύμφωνο σταθερότητος χάνει την αξιοπιστία του όταν λαμβάνονται μέτρα άνισα. Χρειάζεται λιγότερος αυτόματος και ομοιόμορφος χαρακτήρας στην εφαρμογή του συμφώνου γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος ώστε να εξισορροπηθούν μακροπρόθεσμα τα δημοσιονομικά όλων των χωρών της Ένωσης. Στόχος του Συμβόνου ήταν η πρόληψη και η επιτήρηση πολυμερός των ελλημάτων μέσω ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Στο πνεύμα της έκθεσης Συκλούνα νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε την υγεία αυτού του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπηρεσίας για την προειδοποίηση συστημικών κινδύνων γιατί η δημοσιονομική και οικονομική κρίση πρέπει να μας οδηγήσει στη δημιουργία νέων μηχανισμών αμοιβαία αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μελών και ενδυνάμωση των εργαλείων συντονισμού για να υπάρξει μια κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Η κρίση μας δείχνει ότι χρειαζέται περισσότερη δημοσιονομική και φορολογική ευθύνη και περισσότερη επιτήρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ Σίλε για Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Αλμούνια μας είχε πει στο Στρασβούργο πως εάν δεν συμβεί τίποτα το εξαιρετικό η Εστονία θα μπει το 2011 στην Ευρωζώνη. Άλλαξαν τα πράγματα όμως και στην Εστονία και στην Ευρωζώνη. Η Εστονία είναι κατ' ουσίαν η μόνη χώρα της Ένωσης που εκπληρώνει τα κριτήρια του Μάστριχ. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν εάν δεν μπαίνουμε στην Ευρωζώνη. Είναι δηλαδή τόσο χάλια η Ευρωζώνη που δεν μπορεί να αφήσει να μπει μία μικρή αλλά αξιόπιστη χώρα ε, στην Ευρωζώνη. Έχουμε κρεμάσει δηλαδή στην πόρτα της Ευρωζώνης μία πινακίδα κλειστό λόγω ανακαινήσεως. Πήγαμε εμεί στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, λάβαμε σκληρά μέτρα, μειώσαμε το έλλειμμα του ΑΕΠ, είχαμε ανεργία, γιατί λοιπόν ε, να τα κάνουμε όλα αυτά για να πληρώσουμε τα χρέη, τα ιδιωτικά χρέη και όλες χωρών που μπήκαν στο ευρώ. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Νταβίτ Κάζα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το 2008 ήταν πολύ σημαντικό έτος για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Ήταν ε, έτος μεγάλης αβεβαιότητας όσον αφορά την έκταση της κρίσης που μόνο χειροτέρευε. Βεβαιότητα και ε, για το πόσο θα χρειαζόταν να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία και για το ποια εργαλεία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για την ανάκαμψη. Άρα ήταν μια χρονιά δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είχε πολλές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του 2008 συνεννοήθηκε και με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες η ΕΚΤ για να δώσει μια συντονισμένη απάντηση με βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. Η προσέγγιση αυτή της ΕΚΤ αποδείχτηκε πολύ επιτυχής. Πρέπει να υποστηρίξω τον συνάδελφο λοιπόν όσον αφορά τα συμπεράσματά του για την απόδοση της ΕΚΤ. Συμφωνώ πως το 2008 ήταν κέριο και πως οι υπευθυνοί άρχισαν στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, συμφωνώ επίσης με το ότι η μείωση των επιτοκίων δεν πέρασε στους καταναλωτές. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Σημειώστε το λοιπόν κύριε Τρισέ. Συνολικά θεωρώ πως η έκθεση είναι ισορροπημένη, εξαίρετη, όπως ε, την συνέταξε ο συνάδελφος ο Μαλτέζος, ο κύριος Τσικλούνας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Περβάνς Μπερές. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το χρονοδιάγραμμα εμπόδισε τον ε, κύριο Γιούνκερ να είναι παρόν. Έχουμε δύο πολύ καλές εκθέσεις και ε, να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στη συζήτησή μας σε μια κριτική φάση του ευρώ. Η έκθεση Σικλώνα μας επιτρέπει να βάλουμε τη βάση της συζήτησης κυρίως ε, για τους όρους διορισμού της, του διαδόχου σας κύριε Τρισέ, δηλαδή από, από άποψη δημοκρατίας, για τον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας, τη διαχείρισή της. Η έκθεση του κυρίου Γκίγκελ αφορά σε θέματα που εμπίπτουν στη δική σας ε, αρμοδιότητας το ρίσκο της ζώνης ευρώ είναι να αποδυναμωθεί το κοινωνικό μας μοντέλο. Όταν ο κύριος Αλμούνια, ο προκάτοχός σας κύριε Ρεν, έθεσε το θέμα επιτάπητος, μίλησε για κάτι το κραυγαλαίο, την όξυνση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Να που βρισκόμαστε. Και αυτό που οι συντάκτες της συνθήκης και του συμφώνου σταθερότητας είχαν υποτιμήσει. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό για δύο λόγους. Το σύμφωνο σταθερότητας είναι ένα σημείο κλειδί για τα δημοσιονομικά, αλλά είναι ανεπαρκές. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν, δεν έχουν έφεση προς την κύρωση ε, και άρα δεν έχουν και μεγάλη όρεξη συνεργασίας. Πρέπει να βρείτε εσείς λοιπόν το μαγικό ραβδάκι που θα οδηγήσει σε αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να προχωρήσουμε στη φορολογική εναρμόνιση και η έκθεση 20. 20 δεν αναφέρει καθόλου αυτό το σημείο για την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων που πρέπει να συνεχιστεί. Ο κύριος Εσάγια. Κυρία Εσάγια, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα της κρίσης στα δημόσια οικονομικά προκαλούν προβλήματα σε πολλές χώρες και μειώνουν τις κοινωνικές παροχές. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει πρόθεσμα με τα δημόσια οικονομικά. Έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας δυστυχώς οι χώρες δεν το εφάρμοσαν οπότε ε, μένουμε με τα ελλείμματα. Βεβαίως η ουσία του προβλήματος είναι η οικονομική πολιτική Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την απασχόληση και αυτό σημαίνει πως πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις. Πρέπει να ισορροπήσουμε τις δαπάνες, να δούμε τι θα γίνει και με τη βιωσιμότητα και βεβαίως όσο περισσότερο αυξάνονται οι φόροι μακροπρόθεσμα θα υπάρχει μια βάση για τα δημόσια οικονομικά. Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και το πώς αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η συντάξει, η σταθερότητα και η ανάπτυξη είναι σημαντικές, η ανεργία επίσης πρέπει να λάβουμε μέτρα για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και άμεσα βραχυπρόθεσμα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα δημόσια οικονομικά και να έχουμε ισορροπημένους, ε, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν από τον κύριο Ρεν τι σκοπεύει να κάνει για τον συντονισμό των οικονομικών αποφάσεων εν καιρό κρίσης. Πώς οι οικονομίες των κρατών μελών θα ελεγχθούν. Χρειαζόμαστε σφιχτή πολιτική προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Λούντβιχσον. Ευχαριστώ. Τρία βασικά σημεία θέλω να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τα δημόσια οικονομικά Αλλά όχι μόνο οικονομίες. Πώς θα καταπολεμήσουμε και την ανεργία και θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Γιατί εντάξει, σε πολλές χώρες χρειάζονται περικοπές στο δημόσιο τομέα, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθούν τα έσοδα μέσω ανάπτυξης. Να έχουν περισσότεροι άνθρωποι δουλειά και να πληρώνουν φόρους. Στην έκθεση ε, τίθεται το ερώτημα της διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εκεί υπάρχουν πολλά να γίνουν. Η διαφάνεια είναι μια καλή δυνατότητα για να εμποδίσουμε τις επικίνδυνες αυτές συμπεριφορές και ταυτόχρονα σημαίνει πως η επιτήρηση θα είναι πιο αποτελεσματική και άρα θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν πρέπει να παίξει εδώ πέρα ένα ρόλο πρώτο πόρο και να βελτιώσει τη διαφάνεια στις εργασίες της. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν είναι να δημοσιεύει τα πρακτικά του Συμβουλίου της. Χρειάζεται αυτή η διαφάνεια ως βασική αρχή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα οι συστάσεις για τις χώρες ε, που διατρέχουν ιδιαίτερου κινδύνου είναι επίσης αναγκαίες και αυτό ξεκαθαρίζει και στην έκθεση δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι σε καιρούς κρίση να έχουμε σαφή ε, πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα χρειάζεται μια πράσινη στροφή της πολιτικής και Πρέπει να επικεντρωθούμε και στις ΑΠΕΣ, σε νέα συστήματα συγκοινωνιών και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε η φόρο ανάπτυξη. Κυρία Έγκελ. Το 2009 είναι η πιο δύσκολη χρονιά και η πιο χρήσιμη για το ευρώ από τη θέσπιση του διότι είχαμε μια ανταγωνιστική υποτίμηση με φόντο την κρίση και υπέσκαψε και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης. Τίποτα δεν έμεινε απ' έξω από την κρίση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, θέλουμε μια πιο ορατή, πιο έντονη διαφάνεια για το ευρώ. Μόνο η αλληλεγγύη μπορεί να σταματήσει το κερδοσκοπικό κίνημα το οποίο ε, επιτίθεται στην Ελλάδα. Χρειάζεται λοιπόν αλληλεγγύη και η αλληλεγγύη είναι συνώνυμη με τη σταθερότητα. Οι, τα, οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν έβλαψαν μόνο την Ελλάδα, έβλαψαν και το ευρώ χρειάζεται να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας για να αποφεύγουμε τα διέξοδα τα οποία δεν, στο οποία πέφτουν πολλές χώρες την ίδια στιγμή. Χρειάζεται δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου. Γιατί λοιπόν ο πρόεδρος της Ευρωζώνης να μην συμμετέχει στο G20 τις νέες χώρες στην Ευρωζώνη πρέπει να τις υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό και όχι με καχυποψία. Η, η διεύρυνση της Ευρωζώνης πρέπει να συνοδεύεται και με άλλα μέτρα εναρμόνιση των οικονομικών και φορολογικών πολιτικών. Έτσι θα έχουμε και απόλυτη επιτυχία του ευρώ. Σικέρσκι. Πρόεδρε, το θέμα σε περίπτωση κρίσης είναι όχι μόνο η πρόληψη αλλά και η θεραπεία. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει και σε περιπλοκές και σε χειροτέρεψη της αρχικής ασθενείας. Ας δούμε ποιος είναι ο λόγος της κρίσης αυτής. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αμέλεια ή πρόκειται για εξωτερικούς λόγους. Ο, η κρίση είναι μια επίθεση κατά των μηχανισμών της αγοράς. Πρέπει λοιπόν η κερδοσκοπία των αγορών να περιοριστεί για να υπάρξει μεγαλύτερη επιτήρηση των αγορών, ιδιαίτερα όταν παρατηρούνται ασυνήθιστα φαινόμενα. Μέχρι τώρα η επιτήρηση γινόταν από εθνικά κρατικά σώματα ενώ η παγκοσμιοποίηση απαιτεί τη δημιουργία και παγκοσμίων ε, οργανισμών επιτήρησης τουλάχιστον σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο πράγμα το οποίο δεν έχει ακόμα υπάρξει. Μια αγορά βασίζεται σε ορισμένες αξίες Η κρίση που ξέσπασε πέρυσι βέβαια είχε τις ρίζες της ένα χρόνο νωρίτερα και θα μπορούσε να είχε ελεγχθεί από με πολιτικά μέσα και μέτρα. Οφείλεται στην μη επιβολή των ε, συστάσεων που είχαν ήδη γίνει γιατί ορισμένες χώρες ήθελαν να αυξήσουν τα κέρδη τους στην κερδοσκοπία τους μάλλον. Εδώ το πρόβλημα που τίθεται είναι πώς γίνεται η οικονομική διακυβέρνηση. Ενώ μια ένωση σαν τη δική μας πρέπει να έχει κάποια κοινά εργαλεία και επιτήρησης και διακυβέρνησης καθώς και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δεν πρέπει βέβαια να επιβαρύνουμε τους ασθενέστερους πάντοτε με το βάρος της αντιμετώπισης της κρίσης το μελλοντικό, η μελλοντική αυτή υπηρεσία... Όχι, παρα, τελείωσε ο χρόνος σας. Τώρα ο Ότμαρ Καράς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Τρισέ, να σας ευχαριστήσω, όχι για τα τελευταία χρόνια, αλλά για τις τελευταίες εβδομάδες. Ικανός, ανεξάρτητος, συνεπής, εσείς και οι συναδελφοί σας ήσασταν βράχος σταθερότητας. Κύριε Ρεν, οι δηλώσει στις τελευταίες μέρες ήταν ενθαρρυντικέ. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ακολουθήσουμε συνεπώς το δρόμο που χαράξατε. Το ευρώ είναι άγκυρα σταθερότητα και σε καιρού κρίσης και πρέπει να σταματήσουν οι θρύλοι, οι μύθοι εδώ πέρα. Πω το ευρώ και το σύμφωνο σταθερότητα είναι η αιτία των προβλημάτων τη Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργό ο Έλληνα την προηγούμενη εβδομάδα μα είπε δεν φταίει το ευρώ, το ευρώ είναι η λύση. Χωρί το ευρώ δεν υπάρχει μεταρρύθμιση, χωρί το ευρώ δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου. Μην αποδυναμωνόμαστε από μόνοι μας εδώ πέρα. Όταν ήδη η Ελλάδα αισθάνεται προστατευμένη, η Ελλάδα δεν ζητιανεύει λεφτά όπως λένε κάποιες εφημερίδες. Καλό είναι κάποια μέλη του Συμβουλίου έτσι για τον εσωτερικό τους λαϊκισμό να μην κάνουν τέτοιες δηλώσεις, να αναζητήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Δεν ζητάνε λεφτά και δεν μπορούν να λάβουν και τέτοια επιδότηση. Θα είναι μια στήριξη για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού σχεδίου και των οικονομιών που κάνουν. Εδώ πέρα λοιπόν η ΕΚΤ και ο κύριος Τρισέ είπαν με το σχέδιο αυτό των τριών φάσεων πότε είναι δυνατό να γίνει το οτιδήποτε. Και τελειών. Έχουμε νομισματική ένωση αλλά όχι οικονομική ένωση. Για την Οικονομική Ένωση χρειάζεται πολιτική βούληση των κρατών μελών και όχι συμβουλές. Σημαίνει συντονισμός των προϋπολογισμών, φορολογικός εναρμονισμός και συντονισμός και στην κοινωνική και οικονομική πολιτική και στην εκπαίδευση. Αυτή τη δέσμευση αναμένουμε, προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε και προς το συμφέρον του ευρώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάρας. Η κυρία Γιάσλοβιέτσκα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη για τη ζώνη ευρώ. Μπήκε μεν η Σλοβακία στην Ευρωζώνη, αλλά κλείσαμε με την ε, κρίση της Ελλάδας συν την παγκόσμια κρίση. Πώς να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, τι προσανατολισμό πρέπει να δώσουμε στην παγκόσμια οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το ψήφισμα εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο της συζήτησης. Κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση, τα προβλήματα της Ελλάδας, οι συζητήσεις για τη βοήθεια που πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η κατάσταση αλλάζει βαθιά. Ο πρόεδρος Μπαρόσο θέλησε να υποστηρίξει την παροχή ενισχύσεων στις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν προβλήματα αλλά αυτά πρέπει να οριστούν από τα μέλη της Ευρωζώνης. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τη θέση του κυρίου Λεβαντόφσκι και θέλω να υποστηρίξω και τη θέση του κυρίου Ροφστόσκη του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας ενώνω και εγώ τη φωνή μου σε αυτές τις εκκλήσεις όλα τα κράτη-μέλη ακόμη και αυτά που δεν είναι στην Ευρωζώνη θα πρέπει να πράττουν ούτως να ενισχύουν την Ευρωζώνη και η Πολωνία η οποία ακόμη δεν είναι στην Ευρωζώνη θα γίνει και αυτή μέλος της και θα θέλαμε από τώρα να ε, φανταστούμε το μέλλον της Ευρωζώνης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτές τις χώρες από τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να έχουμε μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Δεν μπορούμε να έχουμε μία διάσταση μεταξύ των χωρών Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης. Είμαστε μία ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση στην Κομισιόν και στην Κεντρική Τράπεζα για να διευρυνθεί η ζώνη ευρώ με τα τωρινά κριτήρια και στον πρόεδρο της Κεντρικής ε, Τράπεζας, τον κύριο Τρισέ, τον ευχαριστώ για τη δουλειά του αυτή την τόσο δύσκολη χρονιά. Προχωράμε στο Catch the Eye. Ο συνάδελφος Μεζάρος. Ε, ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές, τον Επίτροπο, τον κύριο Τρισέ που αντιμετώπισαν αυτό το θέμα το τόσο σημαντικό για μας με ιδιαίτερο άνοιγμα πνεύματος και ακρίβεια. Το δημόσιο χρέος και ανεργία συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλες τις χώρες και η Σλοβακία δεν αποτελεί εξαίρεση. Mm. 16% έχει φτάσει η ανεργία στη χώρα μου. Η χώρα μου μόλις μπήκε στην ζώνη ευρώ και αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος βλέπει με καλό μάτι το ευρώ ακόμη και σήμερα είναι σημαντικό για μας το ευρώ να παραμείνει δυνατό να διατηρήσει το πρεστής του η Κομισιόν και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να φροντίσουν γι' αυτό ώστε να μην αποτύχουμε. Χρειάζεται να έχουμε μία κατάλληλη ενσωμάτωση σε αυτό το επίπεδο. Ρίγμαντας μπάζι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λόγω της κρίσης Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δικαιολογημένα τα διάφορα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης τα οποία όμως δεν έχουν εναρμονιστεί μεταξύ τους, δεν έχουν τύχει εναρμόνισης μεταξύ τους. Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματα της έλλειψης αυτής συντονισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν όλο και περισσότερο γιατί δεν στηρίζονται από τις τράπεζες. Η ΕΚΤ έχει κάνει προσπάθειες να στηρίξει τις μεγάλες τράπεζες αλλά για να υπάρξει ίση μεταχείριση πρέπει να υπάρξει και ένας κοινό στόχος ταχείας αναθέρμανσης. Θα έπρεπε η ΕΚΤ να είχε χορηγήσει κεφάλαια και εκτός της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ρεν, όχι, Μπρόνς, Μπρόνς, Μπαλτσάιτης. Ο εισηγητής κύριος Τσικλούνας είπε ότι η ΕΚΤ προσπάθησε να χορηγήσει κεφάλαια αλλά δεν τα πέρασαν οι τράπεζες στους πελάτες των. Το κόμμα μου χαίρεται γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έξω από την Ευρωζώνη γιατί πρέπει μια χώρα να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ίδιας χώρας και όχι στο μέσο όρο των αναγκών 27 χωρών. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε, οι εμπορικέ τράπεζε δηλαδή, χειρίζονται την κυκλοφορία του κεφαλαίου αυτή τη στιγμή. Οι δανειοδοτήσει και η δημιουργία χρήματο πρέπει να φύγουν από τα χέρια των ιδιωτών. Χρειάζονται με περισσότερες δυνατότητες για τους καταναλωτές για να χρηματοδοτούν υποδομές κτλ. Τα τέτοια μεγάλα σχέδια πρέπει να χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και όχι από ιδιωτικές τράπεζες γιατί έτσι ενισχύεται η κερδοσκοπία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκαν. Πρόεδρε οι διακυμάνσεις οι οποίες δημιουργούνται από τα διαφορετικά επιτόκια και από τις ισοτιμίες των νομισμάτων είναι κάτι το οποίο είχαμε βιώσει παλιά, αλλά τώρα η ασπίδα την οποία προσφέρει το ευρώ είναι μοναδικές. Τα πλεονεκτήματα τα οποία προφέρει είναι πράγματι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να παραδεχθούμε μπορέσαμε νομίζω και οι υπόλοιπες χώρες οι εκτός ευρώ να αποφύγουμε τις υπερβολικές διακυμάνσεις ακριβώς λόγω της ύπαρξης του ευρώ. Θα πρέπει και οι οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα ακολουθηθούν από τις ε, υποψήφιες χώρες μέλη για το ευρώ να συνεχιστούν και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την διεύρυνση της ζώνης ευρώ για να μπορέσουμε να προστατευτούμε καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κατόπιν έχει τον λόγο κύριε Κάνη Κάτμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρισέ. Σας ευχαριστώ για το κομμάτι εκείνο της έκθεσης το οποίο προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να μειώσουμε πολύ τους μισθούς. Σας ευχαριστώ γιατί πράγματι έτσι δεν θα βοηθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αλλά δυσκολεύει τη ζωή των Ευρωπαίων εργαζομένων και όσο είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε τους προϋπολογισμούς μας σωστά τόσο σημαντικό είναι να του διαμορφώσουμε και κοινωνικά. Αν έχουμε μια Ευρώπη στην οποία δεν επενδύουμε στην εκπαίδευση, δεν επενδύουμε στην υγεία, στην έρευνα, τότε δεν έχουμε και Ευρώπη ανταγωνιστική και σταθερή. Δεν μπορεί να την πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε για την κρίση. Αν δεν επενδύουμε στους ανθρώπους δεν θα έχουμε μέλλον ως Ευρώπη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην ε, συνθλιβούν τελείως οι κοινωνικές πτυχές. Σας ευχαριστώ και Σόλταν κατόπιν τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησα αμέσως ε, τον λόγο. Έλαβε άλλος συνάδελφος τον λόγο, αλλά σας ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, ως τελευταίος ομιλητής. η κυρία Αγγέλικα Βέτ. Σας ευχαριστώ. Η κρίση αυτή μας αναγκάζει να δούμε τι θα γίνει με τους προϋπολογισμούς και η παγκοσμιοποίηση μας αναγκάζει να παίξουμε έναν ουσιαστικό ρόλο στους προϋπολογισμούς. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει στην πλάτη των απλών ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να είμαστε υπεύθυνοι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνουν λοιπόν εδώ πέρα οι παρεμβάσεις αυτές και τον λόγο έχει ο κύριος Ζανκλώτρης. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Σας κατευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εδώ και 6,5 χρόνια προσέρχομαι τακτικά στο Κοινοβούλιο και για πρώτη φορά βλέπω να έχουν γίνει τόσες αναλύσεις, τόσες προτάσεις, τόσες συστάσεις. Έχω εντυπωσιαστεί από τον πλούτο αυτόν που άκουσα και από τις διάφορες απόψεις που έχουν ακουστεί, από διαφορά των απόψεων μάλλον. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσα απεκόμισα από αυτά που άκουσα που ήταν όλα ενδιαφέροντα, όλα ανεξαιρέτως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τα εκμεταλλευτεί δεόντως. Πρώτον, στη γλώσσα του Νίξον. Θα ήθελα να πω πως ε, αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις και ακούσαμε βέβαια και επένους για το ότι αντέδρασε γρήγορα σε καιρούς δύσκολους. Να σας πω πως θεωρώ πως εγώ και οι συναδελφοί μου κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σε εξαιρετικές συνθήκες, οι χειρότερες από το Δεύτερο Παγκόσμιο και ίσως και από τον Πρώτο Παγκόσμιο. Θα ήταν χειρότερες από τον Παγκόσμιο αν δεν είχαμε δράσει. Και πολλοί είπατε πως οι προκλήσεις ε, υπήρχαν και για άλλες κεντρικές τράπεζες ε, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όλοι λοιπόν πρέπει να αναλάβουμε τις τεράστιες ευθύνε μας και συμφωνώ πλήρως με όσους είπαν πως δεν μπορούμε να πούμε πως πέρασαν τα δύσκολα. Δεν έχουν περάσει τα δύσκολα. Δεν επιστρέψαμε στα φυσιολογικά. Πρέπει να παραμείνουμε σε γρήγορση. Επίσης, έλαβα το μήνυμα για δουλειές και ανάπτυξη. Συμφωνώ με το να έχουμε σταθερότητα, με το να είμαστε αξιόπιστοι μέσω μακροπρόθεσμα, συνεισφέρουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά ξέρετε ότι το μήνυμά μας είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να συνεχιστεί η δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Σημαντικό μήνυμα που έρχεται από εσά και συμφωνούμε με αυτό στην έκτη θέλω τώρα να απαντήσω και εξ ονόματος του Επιτρόπου. Ε, είναι για αυτό για την διακυβέρνηση της Ευρώπης των 27 και των 16 της Ευρωζώνης. Είναι ουσιαστική σημασίας και εμείς είμαστε οι τελικά υπεύθυνοι για τις χώρες και καλούμε τους υπευθύνους ε, να αναλάβουν και εκείνοι τις ευθύνες τους στις χώρες και να επιτηρήσουν. Χρειάζεται πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη, επιτήρηση των ε, δημοσιονομικών πολιτικών που είναι η καρδιά της ΟΝΕ και βεβαίως και επιτήρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των διαφόρων οικονομιών, ειδικά στην Ευρωζώνη. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ άλλο για την Ελλάδα και τα διάφορα ζητήματα που διακυβεύονται. Είχα την ευκαιρία να απαντήσω πολλές φορές στην Επιτροπή, την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Να πω μόνο το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό λέγεται Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα, το είπε κάποιος βουλευτής εδώ πέρα. Και ένα... πήρε πολύ στα σοβαρά το πρόβλημα αυτό, εξάντε με μεγάλη αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και ικανότητες και αυτό το αναγνώρισαν όλοι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η κρίση της ΕΚΤ για τα νέα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση είναι πως είναι πιστικά και θα προσέφτα θαραλέα. Μία κουβέντα για την κατάσταση τη μακροπρόθεσμη στη ζώνη του ευρώ. Τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια θα έχουμε και θα δώσουμε αυτή την σταθερότητα των τιμών όπως την παρήχαμε μέχρι τώρα. Αυτά είναι γεγονότα, νούμερα, δεν είναι θεωρίες. Και επιμένω σε αυτό. Όλα τα μέλη της ζώνης ευρώ γνωρίζουν ότι ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη ευρώ θα είναι κοντά στο 2% ε, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλουν τα κατάλληλα συμπεράσματα για την εθνική τους περίπτωση εποφελούνται από τη συμμετοχή στη ζώνη ευρώ, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική κατάσταση σε επίπεδο πληθωρισμού που θα είναι διαφορετική από αυτό το οποίο εμείς δίδουμε σαν εγγύηση. Το κάνουμε γιατί αυτό μας ζητήθηκε και εμείς παραμένουμε πιστοί στην εντολή μας και είναι κάτι που συνεισφέρει στη σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη. Να κλείσω κύριε Πρόεδρε με δύο λέξεις μόνο. Για το θέμα της διαφάνειας όπως σας έχω ήδη πει και εδώ στα μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε οι πλέον διαφανείς σε όλον τον κόσμο σχετικά με την άμεση δημοσίευση των αναλύσεών μας. Τα statement που εκδίδει η τράπεζα. Αμέσως μετά από το Συμβούλιο των Δικητών Τραπεζών ε, κάνουμε μια συνέντευξη ενημερωτική και το μόνο σημείο στο οποίο δεν αποφασίζουμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις ε, να κάνουμε είναι ότι δεν ανακοινώνουμε το ποιος ψήφισε τι κάθε φορά. Και αυτό ε, το κάνουμε γιατί εμείς δεν είμαστε μια συλλογή ε, μεμονωμένων, λειτουργούμε συλλογικά όμως Είμαστε μια ενότητα και ακριβώς αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζεται σαν Διοικητικό Συμβούλιο και όχι σε επίπεδο μεμονωμένων μελών. Λοιπόν, τα πράγματα είναι έκτακτα και θα πρέπει εμείς όχι μόνο να τροποποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της πληματαγορές, αλλά θα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε για να μην βιώσουμε ξανά στο μέλλον τέτοιου είδους κρίσεις με τις οποίες έπρεπε να ασχοληθούμε μέχρι τώρα. Τώρα για την Πολωνία και την Ουγγαρία. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Μας είπαν ότι δεν τις μεταχειριστήκαμε όπως θα έπρεπε σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω ότι δεν είσαστε σωστά πληροφορημένοι. Θα ήθελα να ζητήσω από την βουλευτή, η οποία έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, να πάρει πληροφορίες από τις κεντρικές τράπεζες των δύο συγκεκριμένων χωρών και θα έχει πλέον τις αποδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις δύο αυτές χώρες προς όφελος της Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Όλυ Ρέν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τη σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση. Άκουσα προσεκτικά τις απόψεις σας. Συμπεραίνω πως υπάρχει ισχυρή στήριξη για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου η σημερινή συζήτηση ε, έστησε το σκηνικό για το Συμβούλιο σήμερα και αύριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θετικό είναι επίσης ότι θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να συνεχίσουμε τη συζήτηση περί οικονομικής διακυβέρνησης στην αρμόδια επιτροπή σας μετά το Πάσχα ε, και ελπίζω σύντομα να έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν δύο πτυχές ε, ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα, ο θεμέλιος λίθος θα είναι αξιόπιστη και πιο προληπτική δημοσιονομική επιτήρηση του προϋπολογισμού και όταν χρειάζεται θα απευθύνονται και προειδοποιήσει στα κράτη-μέλη. Δεύτερο στοιχείο θα είναι πιο αποτελεσματική, συστηματική και έντονη επιτήρηση μακροοικονομικών ανισορροπιών και αποκλήσεων ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Και της ε, Ένωσης και όσον αφορά τώρα τις δεσμευτικές συστάσεις. Αυτές χρειάζονται για να μην σορευτούν ανισορροπίες. Και είναι προφανές πως ε, πιο πιεστική ανάγκη βρίσκεται βέβαια στις χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα και τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ξεκινώντας από την Ελλάδα. Uh, είναι επίσης προφανές πως δεν μπορούμε και δεν πρόκειται με αυτό να εννοήσουμε πως ε, θα μειωθεί η εξαγωγική ικανότητα πλεονασματικών χωρών με πλεονασματικό σύγκεντρο των συναλλαγών. Με άλλα λόγια, στόχος δεν είναι ανα... δεν είναι ανάγκη να κάνουμε την Bayern Μονάχου να παίξει χειρότερα εναντίον ε, της Λιών αλλά να αυξήσουμε την δυνατότητα εξαγωγών όπου χρειάζεται και την εσωτερική ζήτηση έτσι ώστε και η Bayern και η Λιών να παίξουν καλύτερα ως ευρωπαϊκές ομάδες έτσι ώστε και η επίθεση της Bayern και της Λιόν να γίνουν καλύτερες και η άμυνα Αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες, αυτό είναι το νόημα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους. Θα δώσω το λόγο τώρα στους δύο εισηγητές σύντομα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Πρώτος ο κύριος Κυκλούνα. Τρία λεπτά, όχι περισσότερο παρακαλώ. Και θα ήθελα να σας ζητήσω επίσης να μην κάνετε θόρυβο γιατί δεν σας ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα σημεία θα ήθελα να θίξω. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί πράγματι απάντησε στις ερωτήσεις τις οποίες έθεσα και εγώ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές να θυμίσω ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας σε αρκετές ε, από τις τροπολογίες και γι' αυτό υπήρξε αυτή η ε, συζήτηση παραγωγική. Οι εντάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι καινούργιες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν βρισκόμαστε στην βέλτιστη δυνατή κατάσταση σε αυτή τη φάση. Παρόλα αυτά θα πρέπει να φανούμε αισιόδοξοι, θα πρέπει να φανούμε δραστήριοι και νοτόμοι και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οικονομικές αρχές οι οποίες να μην αγνοούν την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Συνοχή. Πολλοί είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα γιατί αυτό απαγορεύεται από την ρήτρα του άρθρου 103 της συνθήκης. Το ακούσαμε αυτό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το να υπάρξει μια ρήτρα σε εισαγωγικά σωτηρίας είναι ένα πράγμα. Αλλά το να βοηθήσει κανείς προσωρινά συγκυριακά θα έλεγα είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες παρέμβασης, κάποιες από αυτές είναι βραχυπρόθεσμες, κάποιες είναι μέσο-μακροπρόθεσμες. Πολλοί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους εξέφρασαν την επιθυμία και αυτό το συμμεριζόμαστε νομίζω όλοι η Ευρώπη σε κάθε της προσπάθεια να στέφεται από επιτυχία. Αυτό θέλουμε όλοι και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα πρέπει εν πάση περιπτώσει να καταλήξουν σε μια λύση που θα μας οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Και θα πρέπει φυσικά κάνοντας το αυτό να ξεπεράσουμε κάποιες επιφυλάξεις οι οποίες υπάρχουν εναντίον και εις βάρος αυτή τη στιγμή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του ρόλου τους. Θα πρέπει τέτοιου είδους κρίσεις να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ τον κύριο Σκυκλούνα. Θα δώσω τον λόγο στον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Γκίγκολντ. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Κύριε Γκίγκολντ, δύο λεπτά. Μετά από τη συζήτηση αυτή, να μου επιτρέψετε να σημειώσω ε, τρία πράγματα. Πρώτον, ακούσαμε πολλές φορές διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει ομοφωνία σε σχέση με αυτές τις, ε, με αυτές τις ενδείξεις έλλειψης ισορροπίας που χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ προς τους κυρίους κυρίους ε, Τρισσέ και να μην είσαστε ημίτυφλοι στον τρόπο που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Έχουμε υποτίθεται συμφωνήσει επί της ουσίας ότι τα κόστη θα αυξηθούν σε σχέση με τους στόχους που έχουμε στον τομέα του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας και κάποιες χώρες ξεπέρασαν τα όρια και καλά κάνετε και ε, παρεμβαίνετε. Υπάρχουν άλλες χώρες όμως οι οποίες χρησιμοποιούν τη φορολογική τους πολιτική για να παραμένουν κάτω από τα ποσοστά αυτά. Και αν δεν στρέψετε την προσοχή σας και προς αυτές τις χώρες τότε τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα και τότε νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα υπονομεύσουμε σαφέστατα τα οικονομικά θεμέλια της Ευρωζώνης. Παρακαλώ ανοίξτε και το άλλο μάτι. Ζητώ και από τους συναδέλφους επίσης να κάνουν το ίδιο. Ας κοιτάξει κανείς το ελληνικό παράδειγμα και ας κοιτάξει το πρόγραμμα σταθερότητας. Να υπογραμμίσω εδώ ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα και αναφέρομαι και στην επίσκεψη που έκανα στην Ελλάδα την προηγούμενη ε, εβδομάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια πάρα πολλοί έγιναν πάρα πολύ πλούσιοι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν χαρακτηριζόντουσαν από δίκαιες ευκαιρίες. Και ναι μεν εσείς πενέψατε την Ιρλανδία αλλά δεν μπορείτε να τη συγκρίνετε με την Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες πιστεύουν ότι πρέπει να υποφέρουν για πράγματα τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν προκαλέσει. Και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ρέν να πιέσετε την ελληνική κυβέρνηση και να αντιμετωπίσει πραγματικά με σοβαρό τρόπο τον παράνομο πλούτο που έχει ισορρευτεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γιατί τότε οι δυσκολίες ε, αν δεν γίνει αυτό θα είναι πάρα πολύ ε, μεγάλες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα ίσως να μην είναι απόλυτα κοινωνικά δίκαια. Ευχαριστούμε και θα ψηφίσουμε σε λίγο. Ιταλίας Ο Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ κύριε. Διότι θα αρχίσει η ψηφοφορία. Για προσωπικό. Έχει στήσει το λόγο κάποιος συνάδελφος. Τρεις μινούτος. Επί προσωπικού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, 19 Μαρτίου, λέει ο κύριος Γκόλνης, δηλώθηκε ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου παραβίασε ένα, μια διάταξη διότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Διεθνούς Πρωτοκόλου για την ασυλία δεν, δεν με προστάτευσε το Κοινοβούλιο επί τη βάση της καταγγελής Ρωμανιόλη. Δηλαδή εγώ υπέστη δίωξη πολιτική, νομική, ε, προσωπική, διότι